Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Πρώτα απ' όλα να σας θυμίσω ή μάλλον να ζητήσω την έγκριση των όσων συζήτησαν και πρότειναν οι συντονιστές χτες. 118-117 έτοιμα ερμηνεία των άρθρων αυτών ε, θα υποβληθεί το αίτημα μέσω επιστολής του Προέδρου σας. Όσον αφορά τον, την νομοθετική πρόταση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, έκθεση Giggold και την έκθεση για, την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, χθες δεν βρεθήκε συμφωνία όσον αφορά την, τον ορισμό δύο, ε, των δύο εισηγητών. Όμως ε, υπήρξε συμφωνία ε, με τον κύριο Γκουαλτιέρη και μπορώ να σας πω ότι ο εισηγητής για την ας πούμε έκθεση Γκίγκολτ θα δοθεί στο ΕΛΚΕΝΟ, η Άλντε θα αναλάβει την έκθεση ε, δηλαδή την γνωμοδότηση σχετικά με την έκθεση Τίσεν. <clears throat> Όσον αφορά νομοθετική πρόταση για τα ιστορικά αρχεία, είναι μια πρόταση με την οποία ασχολούμαι εγώ προσωπικά προτείνουν οι συντονιστές να μην υπάρξει καμία ε, πρόταση όσον αφορά την απαλλαγή για την τροπολογία του 2011 και να μην δοθεί ε, ε, συνέχεια στο θέμα του που υπέβαλε ο κύριος Φοντάνα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Όσον αφορά τώρα ακροάσεις και αποστολές οι συντονιστές προτείνουν να οργανωθεί μία επίσκεψη στα Ηνωμένες Πολιτείες με ένα πολύ καλό προετοιμασμένο πρόγραμμα γιατί έτσι θα είναι και πιο εύκολη η αδειοδότηση αυτής της ε, ε, επίσκεψης. Επίσης, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί τα θέματα τα συνταγματικά είναι πάρα πολύ έντονα και καλό είναι να συνεχίσουμε έναν ικανό διάλογο. Επίσης, μοιράστηκε το πρόγραμμα για την έκθεση στην Ιρλανδία και θα σας δοθούν περαιτέρω πληροφορίες αργότερα. Επετέχθη συμφωνία όσον αφορά ε, τις ε, διασκέψεις καθώς επίσης και τις μελέτες για τον επόμενο χρόνο. Δεν είχαμε χρόνο να μελετήσουμε εντελεχώς το θέμα αυτό. Θα υπάρξει γραπτή διαδικασία. Βάσει σύστασης ε, του εισηγητού κυρίου Νταφ όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 9309 σχετικά με την δυνατότητα να είναι κανείς υποψήφιος σε χώρα διαφορετική από την χώρα διαμονής του αποφασίσαμε η νέα διαβούλευση για το θέμα αυτό να γίνει βάση της ε, απλουστευμένης ε, διαδικασίας ε, που προβλέπεται στο άρθρο 46. Γρήγορη έγκριση χωρίς τροπολογίες επί του κειμένου. Για λόγους ε, Γρηγοράδας ε, θα αποφασιστεί αυτό αμέσως. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω στον ε, συνάδελφο Νταφ να περιγράψει λίγο αυτή την εργασία έτσι ώστε να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Λέω ο κύριος Νταφ. Όπως σωστά είπατε, πρόκειται για την κατάληξη της διεκπαιρέωσης αυτής της έκθεσης που προσπαθήσαμε να την ολοκληρώσουμε ανεπιτυχώς την τελευταία θητεία του Κοινοβουλίου. Ξεκίνησε το 2007 η υπόθεση και οι διαπραγματεύσεις κόλλησαν στο Συμβούλιο αλλά πρόσφατα είχαμε απεμπλοκή του θέματος μια που επιφέραμε κάποιες δευτερεύουσες βελτιώσεις όσον αφορά την διαδικασία της ε, έγκρισης υποψηφιωτήτων στις χώρες πρόλευσης και δεν κατέστη δυνατόν να καλυφθούν όλα όσα θέλει το Κοινοβούλιο αλλά νομίζω ότι συμφώνησαν οι συντονιστές ότι τίποτα καλύτερο δεν μπορούσαμε να πετύχουμε όσον αφορά την πλοκή ε, μεταρρύθμιση πριν ε, υπάρξει κάποια καινούργια συντακτική συνέλευση. Οπότε έχουμε αυτές τις δευτερεύουσες βελτιώσεις. και θα δούμε τι θα κάνουμε μέχρι το 2014 και έχουμε τη διαδικασία του άρθρου 46 οπότε και μέχρι τότε θεωρούμε ότι θα είναι, είναι ο πιο δόκιμος τρόπος. Στην έκθεση θα σχολιάσουμε αυτές τις ε, βελτιώσεις θα την υποβάλουμε αυτή την έκθεση τον Νοέμβριο στην Ολομέλεια. Ωραία, αυτή είναι η πρόταση. Βάσει του άρθρου 46 και αν δεν αντιτίθεται κανείς, εγκρίνεται η ταχεία διαδικασία. Για να σταματήσει αυτό το αίτημα θα πρέπει να υπάρξουν τουλάχιστον τρεις βουλευτές. Δεν νομίζω ότι αντιτίθενται αυτοί οι τρεις βουλευτές, άρα προχωράμε με απλουστευμένη διαδικασία. Δηλαδή θα εγκριθεί χωρίς τροπολογίες το κείμενο που έχει ε, δώσει το Συμβούλιο και θα το μελετήσουμε, θα υποβληθεί μάλλον στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε και προχωράμε τώρα στην ε, κανονική μας ημερήσια διάταξη και βάσει του πρώτου σημείου που είναι βεβαίως το σημείο 11 της συνολικής ημερησίας διατάξεως, όχι 10, 10, 10 διορθώνει ο Πρόεδρος, 10 διορθώνει ο Πρόεδρος. Ah, sì, sì. Vede il tema della, per eh, cui abbiamo nominato i relatori, prego. Λοιπόν, να ορίσουμε τους εισηγητές. Ε, έχετε κάποιο ερώτημα. Αυτό το σχέδιο ψηφίσματος αφορά τη δήλωση Επιτροπής σε σχέση με τις εκλογές. Και συνεφώνησαν οι συντονιστές να απευθυνθούμε στην Επιτροπή για να εκδώσει ακριβώς αυτή την ανακοίνωση. Και Και συντρέχει εδώ η διαδικασία του άρθρου 110. Έχουμε βέβαια στείλει το σχέδιο ψηφίσματος για να του ρίξετε μια ματιά ο κύριος Σεύκοβιτς αργότερα θα έρθει οπότε μπορούμε να το συζητήσουμε μαζί του. Υπάρχουν εδώ τρία στοιχεία σε σχέση με την αλληλεπίδραση των ευρωεκλογών και την, τον ορισμό της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτά θέλω να τα συζητήσουμε. Ευχαριστούμε. Εγώ ήθελα να ε, ε, προτείνω το ερώτημα αυτό για το οποίο συζητήσαμε ε, με τους συντονιστές την παρουσία του Επιτρόπου Σέρκοβιτς. Εσείς το εισήγατε, μπορούμε να το ξαναυποβάλουμε. Και βεβαίως δεν θέλω να αργήσουμε γιατί 10 η ώρα είπαμε ότι θα κάνουμε τις ψηφοφορίες και επομένως να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε και το σημείο 10. Βεβαίως ευχαριστώ τον συνάδελφο για την πρώτη του παρουσίαση που βεβαίως θα ε, παρουσιάσει εκτενέστερα το θέμα ε, όταν θα είναι εδώ ο Επίτροπος τροποποίηση του κανονισμού 109 του 2010 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών όσον αφορά τη διαδραστικότητά του με τον, με, τον άλλον κανονισμό του Συμβουλίου που αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ειδικά καθήκοντα σχετικά με την προληπτική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Θα συζητήσουμε μαζί λοιπόν τις προτάσεις αποφασίσαμε ε, ότι τις δύο σχετικές εκθέσεις θα κάνουν το ALDE και το ΕΛΚ, δεν ξέρουμε όμως ακόμα συγκεκριμένα ονόματα. Ε, πάντως μπορεί κανείς να μπορούμε ήδη να ξεκινήσουμε τη συζήτηση ελεύθερα ε, και αν θέλει κάποιος να πάρει το λόγο παρακαλώ να μην διστάσει. Ο συνάδελφος uh, um, Νομίζω ότι για την Επιτροπή μας το πιο σωστό είναι να πρόβουμε στη σύνταξη έκθεσης για αυτά τα σημαντικά θέματα η Επιτροπή μας σταθερά θα πρέπει να εμένει στο ότι επιβάλλεται η τήρηση της συνθήκης στο βωμό τη συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που αυτό για μας είναι υψηλή προτεραιότητα. Και όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση, υπάρχουν μείζωνα προβλήματα. Και έχουμε τις χώρες που είναι στην Ευρωζώνη, που είναι στην Τραπεζική Ένωση και αυτοί που δεν είναι και εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι η μόνη χώρα η οποία απολάβει αυτής της παρέκκλησης σε σχέση με το νεονόμισμα. Βεβαίω, Βεβαίως. Στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνονται περισσότερες χρηματοπιστωτικές αλλαγές της Ένωσης. Επομένως αυτό αποτελεί πρόβλημα. από πλευρά νομική συνέπεια και πολιτική συνοχή. Επίση, θα πρέπει όντω να υπάρχει ένα υποπτικό μηχανισμό στην ε, Κεντρική Τράπεζα που είναι λογοδοτή, είναι υπόλογο τέλο πάντων σε κοινοβουλιακή συμβούλια και ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία τράπεζα στα θέματα νομισματικής πολιτικής. Η Επιτροπή έχει προτείνει αυτό που λέμε κινέζικο τείχος το οποίο θα συγκροτηθεί στην Φραγκφούρτη. Και αυτό το συνικό τείχος θα διέπεται από την κατανομή αρμοδιοτήτων όπως ορίζονται, προβλέπονται στην Κεντρική Τράπεζα. Άλλο τρίτο στοιχείο είναι το εξής. Η εποπτεία δεν θα καλύπτει τον τομέα των ασφαλιών όμως αυτό είναι αχίλιος πτέρνα στο σύστημα εποπτείας που θέλουμε να υπάρχει. Για όλες τις χρηματοπιστωτικές αλλαγές. Το τέταρτο στοιχείο πρέπει να το εξετάσουμε είναι η σχέση μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και της έκθεσης Kingold. Γιατί η EBA θα συνεχίσει να έχει την αρμοδιότητα του να καταρτίζει ό,τι προβλέπετε για τους 27. Επομένως, αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουμε. Η ΜΠΑ είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Να δούμε επομένως τι εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης υπάρχουν. Ας πούμε θα μπορούσαμε να έχουμε συγχώνευση των ε, υπαρχουσών σήμερα τριών αρχών εποπτείας και έτσι να αναβαθμίσουμε τις αρμοδιότητες του φορέα συστημικού κινδύνου ούτως ώστε να έχουμε γέφυρα μεταξύ Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και της Κεντρικής Τράπεζας. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μια τέτοια εναλλακτική προσέγγιση έχει ληφθεί υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά Αποφασίστηκε στην Οικονομική Επιτροπή να απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Οικονομική Επιτροπή, να απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον κύριο Ντράγκη για να αναζητηθεί το πνεύμα το οποίο διέπει τις ε, προτάσεις τους. Μην κατακλείδη. Πρέπει να τονίσουμε το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ σφιχτό. Το δε Συμβούλιο είπε ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα Χριστούγεννα. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ αφελές. Ε, και εν πάση το κοινοβούλιο θα πρέπει να δείξει αποφασιστικότητα και να διεκπαιρεώσει όσο γίνεται ταχύτερα το θέμα. Αλλά βέβαια, πάνω απ' όλα, επιβάλλεται να έχουμε μια ποιοτική συμφωνία όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση, που θα πρέπει να είναι βιώσιμη και πραγματικά να ωφελεί τον ε, τραπεζικό τομέα σαν κανονιστική αρχή. Οι τραπεζίτες, ξέρετε, είναι ξυπνότεροι, τουλάχιστον πιο διεκπαιρεωτικοί από την ε, δημοκρατική, ας την πούμε έτσι, ή νομική διαδικασία. Αυτό είναι η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρόκληση. Ευχαριστώ πολύ. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Γκερέρο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Ντάφ για την εισήγησή του και ε, στα όσα είπε στο τέλος ο κύριο Ντάφ με βρίσκει σύμφωνο δηλαδή σε σχέση με την βιασύνη με την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι όχι μόνο ε, σημαντικά για σήμερα αλλά είναι κομβικά όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση του μέλλοντος της Ευρώπης και κρίμα επομένως που θα πρέπει να κινηθούμε τόσο βιαστικά, τόσο πιεσμένα. Τέλος πάντων, εμείς κάνουμε ότι πέρα από το χέρι μας, ούτω ώστε να μην μας χρεώσουν εμά την καθυστέρηση για την ε, μη λήψη αποφάσεων για αυτά τα θέματα και όπως όλοι γνωρίζουμε τα τραπεζικά προβλήματα είναι η πηγή, η αιτία της κρίσης η οποία σοδεί εδώ και σχεδόν μια πενταετία οπότε εντάξει ε, άλλαξαν κάπως τα πράγματα στη διαδρομή και η κρίση μεταμορφώθηκε σε κρίση του κρατικού χρέους αλλά τώρα, τώρα εν πάση ξέρουμε ότι σε κάποια κράτη τουλάχιστον όπως και στην Ισπανία υπάρχει θέμα, υπάρχει κρίση τραπεζική αλλού ε, κάπως υποβόσκει το θέμα αυτό αλλά πάντως έτσι ισχύει, όπως και σε κάποιες ε, χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και δεν θα τις κατονομάσω για να μην μου ανταποδώσουν το κομπλιμέντο. Τέλο πάντων. Ξέρετε τι εννοώ. Πρόεδρε, και εσείς από μια τέτοια χώρα προέρχεστε που επιδέχεται τέτοια αντίπεινα. Τέλος πάντων, η διέξοδος από το τούνελ είναι και περνάει μέσα από τη σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα. Και επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το σύμφωνο σταθερότητας του Μαριοντράγκη, ε, εκείνο και το έγγραφο που αφορούσε την ε, αυθεντική ε, νομισματική ένωση, το οποίο το παρουσίασε ο Φαν Ρομπάι, αλλά έχει περάσει και από άλλε σημαντικέ προηγούμενε προεδρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε όλα αυτά τα κείμενα που λέω, ε, τονίζεται το ότι πρέπει να βελτιωθεί, να γίνει πιο ε, κεντροκατευθυνόμενη, πιο συντονισμένη η τραπεζική υποπτία, Γιατί θεωρείται αδιαμφισβήτητο ότι ε, πέραν του ότι είναι ανοιχτέ οι τραπεζικέ αγορέ, Άπαξ και είναι ανοιχτέ αυτέ, άπαξ και έχουμε ολοκλήρωση τραπεζική στην Ένωση. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά, παρόλα αυτά, σε κάποιο μεγάλο βαθμό ή σε άλλο βαθμό 100% η εποπτεία είναι κατατμημένη ανά κράτος μέλος. Οπότε αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι ε, για το μέλλον να δούμε πώς θα έχουμε ολοκλήρωση της τραπεζικής αγοράς και πώς θα έχουμε ταυτόχρονη την εθνική εποπτεία. Άρα να κάτσουμε και να συγκροτήσουμε κάποιους μηχανισμούς εποπτείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση να, από που προέρχονται τα προβλήματα τα οποία μας εξήγησε ο κύριος Νταφ πρώτα-πρώτα. Που είναι προφανές ότι εδώ πέρα δεν είναι θέμα του πώς θα υποκαταστήσουμε τις εθνικές ευρωπαϊκές αρχές, αυτές που ήδη υπάρχουν, που έχουν συγκροτηθεί από την Κεντρική Τράπεζα. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να προσδώσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά του ε, ολοκληρωμένου μηχανισμού εφοπτεία σε επίπεδο Ένωση. Το δεύτερο τώρα πρόβλημα, ε, στο οποίο επίση μα ε, έκανε κοινό ο κ. Ντάφ, είναι το τι θα κάνουμε, πώ θα κινηθούμε σε μια πραγματικότητα κατά την οποία έχουμε 10, 10 χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν μπει στην Ευρωζώνη. Εκεί τα πράγματα είναι κάπως πιο περιπλεγμένα όσον αφορά την ε, Τραπεζική Ένωση. Εκεί κάπως θα τα βρει δύσκολα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης, ε, είναι και το θέμα των ασφαλιών μας είπε ο Ντάφ και εγώ συμφωνώ μαζί του ότι η εποπτεία θα πρέπει γιατί δεν αρκεί να υποπτεύουμε τις τράπεζες και να έχουμε και άλλους μηχανισμούς, κυρίως τα χρηματοπιστωτικά, που να έχουν κάποιες λειτουργίες που επιδέχονται εποπτεία και εποπτεία μάλιστα ολοκληρωμένου χαρακτήρα. Τέλος, θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το οποίο μας είπε ο κύριος Ντάφτο, αυτό το περίφημο συνικό τείχος. Και αναζητεί διέξοδο για να μπορέσει να περάσει από το τείχος. Γίνεται αυτό. Υπάρχουν μηχανισμοί προς το το. Πάντως, να σας πω μια σκέψη μου όσον αφορά αυτούς τους ομόγεντρους κύκλους που θα μπορούσα να πούμε ότι είναι τμήμα αυτού του συνοικού τείχους. Κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη των περισσότερων της πολιτικής μου ομάδας και λέω ότι τους περισσότερους γιατί πάντα κανείς θα πρέπει να επιφυλάσσεται και να περιμένει να δει ποια θα είναι η τελική τοποθέτηση της Οικονομικής Επιτροπής. Λέω εγώ λοιπόν ότι η πλειοψηφία από εμά πρεσβεύουμε το ότι θα πρέπει και η Κεντρική Τράπεζα να υποπτεύει όλε τι τράπεζε, όλου του χρηματοπιστωτικού οργανισμού. Και γι' αυτό και αυτό το, το λέμε ολοκληρωμένη αποπτία. Και ε, ξέρουμε ότι καταρχήν δεν είναι ρεαλιστικό να ισχυριστεί κανείς ότι μπορεί η Κεντρική Τράπεζα να αρχίσει την υποπτία 6.000 τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρύματων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα μπλοκάρισμα σε όλο το σύστημα. Και φυσικά να, να φτάσουμε σε αποτελέσματα αντίθετα των επιδιωκομένων από αυτή την εποπτεία που θέλουμε να αναθέσουμε στην ε, Κεντρική Τράπεζα. Άρα θα πρέπει να προχωρήσουμε βήμα-βήμα προς την υλοποίηση αυτού του πολιτικού μηχανισμού. Να ξεκινήσουμε επομένω από ένα μικρότερο κύκλο ύλη και μετά σιγά σιγά να ανοίξουμε αυτόν τον κύκλο και να φτάσουμε σε αυτό το συγκροτικό μα μας είπε ο Νταφ που θα περιχαρακώσει όλο το σύστημα των τραπεζών στην Ευρώπη. Δεν είναι απλά θέματα αυτά. Δεν είναι διότι, ξέρετε, είμαι αναπληρωτής στην Οικονομική Επιτροπή και εκεί έχω ακούσει τις ίδιες συζητήσεις που αφορούν τη συστημική πλευρά του τραπεζικού τομέα. Πάρα πολύ επομένω θα ήθελαν μόνο οι συστημικές τράπεζες να υποπτεύονται από την κεντρική τράπεζα. Και αυτό όμως θα μπορούσε να ισχύει και όσον αφορά αυτή τη διάσταση της τράπεζας και εκτός από τη διάσταση θα πρέπει να μπορούσε να καλύψει και την διεύρυνση των εργασιών και των αρμοδιοτήτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλέ τράπεζε που οι χρηματοπιστωτικέ του εργασίε γίνονται μόνο σε μία χώρα. Ή υπάρχουν άλλε που είναι μικρότερε, οι οποίε όμω ε, ε, ε, λειτουργούν σε περισσότερε από μία χώρα. Άρα είναι δύσκολο και ο διαχωρισμό, η διάκριση μεταξύ συστημικών και μη τραπεζών. Πάντως όπως έχουν τα πράγματα νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι το ότι η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να είναι αυτό ο οποίο θα εποπτεύει το, το, το κλάδο, το, το, σύστημα το τραπεζικό στην Ευρώπη. Οπότε νομίζω ότι και εμείς και φυσικά η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να δει τι είδου χάρτη πορεία θα πρέπει να φτιάξουμε, ώστε να μπορέσουμε να, να προχωρήσουμε και σιγά σιγά να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Ξεκινάμε λίγο λίγο και, τελικά, και διευρύνουμε τελικά τη δραστηριότητα για να καλύψουμε αυτό που θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σταρκόφσκι. Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί τα περισσότερα ήδη ελέγχθησαν ιδίως από τον Άντριου. Νομίζω ότι ό,τι και να κάνουμε πρέπει καταρχήν να διευκρινίσουμε τη σχέση μεταξύ όλων αυτών των ε, θεσμικών οργάνων. Γιατί αν ε, στη Συνταγματική Επιτροπή ε, επικρατεί σύγχυση για τα καθήκοντα που πρέπει να έχει το κάθε θεσμικό όργανο, φανταστείτε πόσο μπλέκονται όλοι οι υπόλοιποι για αυτές τις πολύπλοκες δομές. Ιδίω διότι έχουμε δημιουργήσει κάποια θεσμικά όργανα το 2010 και μετά κάναμε κάτι σαν να προσπαθούμε να υπονομεύσουμε το ρόλο τους και να τις παρακάμψουμε θέλουμε τώρα αυτά τα όργανα να τα κάνουμε συμβατά και θέλουμε να το κάνουμε με τρόπο ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα των χωρών που είναι μέσα στην Ευρωζώνη και ε, να λάβουμε υπόψη και τις χώρες εκτός Ευρωζώνης που θέλουν να συμμετάσχουν. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε τη σωστή σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό το καθήκον και πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην υπάρχουν στρεβλώσει στην εσωτερική αγορά. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ιδρύθηκε ακριβώς για να παίξει αυτό το ρόλο και νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνατότητες που έχει για να το πράξει. Και για την έκθεση Giggold πρέπει να εξετάσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν να αλλάξουν οι κανόνες ψηφοφορίας, ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να είναι πιο αποτελεσματική για την ενίσχυση ε, των ε, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Και ο Άντριου έθεσε ένα ερώτημα για το κατά πόσο τα μέλη που θέλουν ε, να ενταχθούν στο σύστημα μπορούν να το κάνουν κράτη-μέλη που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης. Κατά πόσο μπορούν να συμπεριλαμβάνονται. Θα, πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να τους συμπεριλάβουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Πρέπει να δούμε ότι δεν πρόκειται μόνο για τις χώρες της Ευρωζώνης και άλλες χώρες θα θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το σύστημα. Όπως συνέβη και με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Συμφωνώ λοιπόν με τους προλαλήσαντες ότι θα πρέπει να εξετάσουμε όλα αυτά τα θέματα λεπτομερώς και το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να δείξουμε ότι το σύστημα που δημιουργήσαμε πραγματικά είναι ένα αξιόπιστο σύστημα και σαφώς περιγράφει τα καθήκοντα και δεν υπάρχει επικάλυψη και δεν αφήνουμε κάποιες ε, γκρίζες ζώνες, ιδιαίτερα όταν θέλουμε να πληροφορήσουμε την κοινή γνώμη. Διότι αν δεν διευκρινίσουμε τους κανόνες, μπορεί να δίνουμε την εντύπωση ότι το σύστημα που δημιουργήσαμε το 2010 υπονομεύεται από τις αποφάσεις του 2012. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λειτουργήσει το σύστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση που κάνουμε σήμερα. Διαβάζοντα αυτό το έγγραφο τη Επιτροπή, ακριβώ αυτό θέλω να δούμε, τι καθήκοντα θα έχει αυτό το όργανο. Εποπτεία της αγοράς ε, είναι σαφές καθήκον, αλλά ποια θα είναι τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, γιατί όλες, ε, όλοι αυτοί οι οργανισμοί πρέπει να έχουν όλα τα πιστοτικά ιδρύματα, πρέπει να έχουν άδεια από τις αρχές για να μπορούν να λειτουργήσουν. Αυτό το καθήκον θα το αναλάβει στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αποφασίζει αν, μια, αν ένα πιστοτικό ίδρυμα εθνικό ή διεθνέ μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τις δραστηριότητές του. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό ερώτημα. Ποιο θα λαμβάνει αυτή την απόφαση. Στο μέλλον θα τη λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε συνεργασία με τι εθνικέ αρχέ ή οι εθνικέ αρχέ θα λαμβάνουν αυτή την απόφαση. Αν τη λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, νομίζω ότι από νομική πλευρά είναι ενδιαφέρον να δούμε αν ε, αυτά συνάδουν προ το άρθρο 127 σημείο 6 τη συνθήκη, που αποτελεί τη βάση για την πρόταση αυτή. Διότι το άρθρο τη συνθήκη μιλάει μόνο για καθήκοντα και ε, όχι για εξουσία, όχι για αρμοδιότητα που λέει ότι μπορούμε να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθήκοντα αλλά όχι εξουσίες και υπάρχει ε, ε, διαφορά μεταξύ των δύο και θα πρέπει η νομική υπηρεσία να διευκρινίσει τι ισχύει στην πράξη με βάση το άρθρο αυτό. Επίσης, είναι πολύ ενδιαφέρον το τι θα γίνει με τις χώρες εκτός Ευρωζώνης. Τι επιπτώσεις θα υπάρχουν και τι επιρροή θα έχουν σε αυτό το νέο όργανο. θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θα συμβεί με το Ηνωμένο Βασίλειο, παραδείγματο χάρη. Όλα θα αποφασίζονται βάσει αυτού του άρθρου και θα πρέπει να γίνονται όλα αυτά ομόφωνα. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη. Δεν ξέρω, ο κύριο ταυτή έχει να, να πει από αυτού. Τι θα ψηφίσουν όμω και πώ θα ψηφίσουν, θα μπλοκάρουν αυτή τη διαδικασία. Από πολιτική πλευράς λοιπόν πώς το βλέπουμε αυτό το θέμα. Τα νομικά ζητήματα όμως είναι τα πιο σημαντικά και πιστεύω ότι το άρθρο 127 σημείο 6 δεν δίνει μια σαφή απάντηση για το αν μπορούμε να αναθέσουμε τέτοιες εξουσίες, τέτοιε αρμοδιότητε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το έγγραφο τη Επιτροπή επίση δεν δίνει σαφή απάντηση, γι' αυτό θα ήθελα να το διευκρινίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νταφ. Πολύ σύντομα. Νομίζω ότι το άρθρο 127 σημείο 6 μιλάει για ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων ε, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μπορεί να υπάρχουν διάφορα καθήκοντα, συγκεκριμένα καθήκοντα. Το εύρος των λειτουργιών λοιπόν μπορεί να ε, είναι πολύ μεγαλύτερο αν ε, χρησιμοποιήσουμε αυτό το άρθρο. Δεν θα πρέπει να το ερμηνεύουμε ως περιοριστική ρήτρα. Αν υπάρχει νομική και πολιτική συμφωνία, θα δούμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μετασχηματιστεί σε κάτι το οποίο δεν είχε προβλεφθεί αρχικά. Τουλάχιστον όχι από την ε, Γερμανική Κεντρική Τράπεζα, την Bundesbank, όταν ε, συντάχθηκε η συνθήκη του Μάστριχτ. Επίσης, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ε, διάφορα μοντέλα κεντρικής τράπεζας τα οποία μπορούμε να εξετάσουμε. Η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, η Τράπεζα της Αγγλίας. Όλα αυτά τα μοντέλα είναι διαφορετικά. Έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες και εξουσίες. Και έχουν και διαφορετική σχέση το καθένα με τις αρχές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Και αν βγαίνει ένα μήνυμα από όλη αυτή την κρίση, αυτό είναι ότι η σχέση μεταξύ των τραπεζών και των ρυθμιστικών αρχών αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Και θα ήθελα εμείς να έχουμε το προβάδισμα, να είμαστε εμείς η προπομπή αυτής της αλλαγής. Και, μισό λεπτό συγγνώμη, να συμπληρώσω κάτι. Για την ερώτηση για τη Βρετανία που έγινε, Νομίζω ότι η τελική απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου θα εξαρτηθεί από την ποιότητα και το περιεχόμενο της εποπτείας που προτείνεται. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τους κανόνες και σε βάθος. Ο κύριο Μέσσερ Σμιτ έχει ζητήσει το λόγο. Πολύ σύντομα για να απαντήσω στον κύριο Νταφ. Πριν από 20 λεπτά νομίζω είπατε ότι εμεί εδώ στην ΑΦΚΟ πρέπει να είμαστε αυτοί που θα ελέγχουν πολύ προσεκτικά την συνθήκη, την εποπτεία τη συνθήκη. και ακριβώ αυτό επικαλούμε και εγώ. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τη, διά, με τη διατύπωση του 127.6, αλλά αυτό που λέω είναι ότι ε, όταν λέει καθήκοντα τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται οι εξουσίε που τώρα συζητάμε και δεν διευκρινίζεται ούτε στην πρόταση της Επιτροπής. Γι' αυτό πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να έχουμε γραπτός μία ερμηνεία του ποιες είναι αυτές οι προβλεπόμενες εξουσίες για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τώρα και τι είδους εξουσίες δόθηκαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο παρελθόν βάσει αυτού του άρθρου για να είναι σίγουρο ότι ε, αυτά που κάνουμε είναι σύμφωνα προς τη συνθήκη και τη διατύπωση. Ε, Ωραία. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συζήτηση για το σημείο 10, αλλά θα πρέπει να καθορίσουμε και το χρονοδιάγραμμα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθόσεις Γκίγκολ και Τάισον θα εγκριθούν την 29η Νοεμβρίου, η γνωμοδότησή μας θα πρέπει να ψηφιστεί ε, στην συνεδρίαση της 27ης Νοεμβρίου. Άρα ε, τρίτη 6 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι λίγη η προθεσμία υποβολής τροπολογιών και για τις δύο προτάσεις. Επίσης, δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι είναι οι θα οριστούν πολύ σύντομα. Θα ζητήσω λοιπόν από αυτούς τους μελλοντικούς ε, εισηγητές ε, να γνωρίζουν αυτές τις προθεσμίες όσον αφορά τις ε, τροπολογίες τους. Λοιπόν, έχουμε πέντε λεπτάκια μέχρι την ώρα της ψηφοφορίας. Ε, ίσως σε αυτά τα πέντε λεπτάκια να δώσουμε τη δυνατότητα ε, στον συνάδελφο Νταφ να παρουσιάσει λίγο πιο σε έκταση την ε, παρουσίαση που έκανε, το θέμα μάλλον που παρουσίασε ε, το πρωί. Αλλά όχι, να μην ξεπεράσουμε την ενδεκάτη. Πολύ σύντομα σας παρακαλώ, ε, κύριε, την δεκάτη, συγγνώμη. Um, Η δήλωση της Επιτροπής για τις εκλογές. Νομίζω ότι υπάρχουν τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι καλούνται τα πολιτικά κόμματα να ορίσουν τους επικεφαλής ε, για μέλλοντες προέδρους της Επιτροπής. Το δεύτερο είναι ότι ζητείτε τουλάχιστον 50% της νέας Επιτροπής να προέρχεται από, το νέο κοινοβούλιο, από τα μέλη που εξελέγησαν το 2014 και υπάρχει προηγούμενο. Ο Μισελ Μπαγνιέ, παραδείγματο χάριν, εξελέγει ευρωβουλευτής και μετά αναβαθμίστηκε, πώ θα το πούμε, μεταφέρθηκε. Λίγους μήνες μετά στην Επιτροπή και έγινε επίτροπο. Νομίζω ότι το 50% από το Συμβούλιο και 50% από το Κοινοβούλιο θα συμβολίζει την ισότιμη τον ισότιμο σχηματισμό ε, ε, του νομοθετικού οργάνου και της Επιτροπής. Ο στόχος και των δύο αυτών προτάσεων είναι να υπάρχει πιο στενή σύνδεση μεταξύ της εκλογικής εκστρατείας του Κοινοβουλίου αφενός και της εκλογής της Επιτροπής αφετέρου. κάτι που έχει σχέση και με το διεθνή κατάλογο, με τη διεθνή λίστα υποψηφίων. Η τρίτη πρόταση έχει σχέση με το πότε θα γίνονται οι εκλογές από τον Ιούνιο, προτείνεται να γίνονται τώρα Μάιο. Ο σκοπός είναι να έχει το Κοινοβούλιο επαρκή χρόνο να οργανωθεί για την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής τον Ιούλιο. Το 2009 χρειάστηκε να το αναβάλουμε, να αναβάλουμε την εκλογή του Προέδρου μέχρι το Σεπτέμβριο και η νέα Επιτροπή δεν μπορούσε να αρχίσει να λειτουργεί μέχρι το Φεβρουάριο. Εξαιρετικά μακρά περίοδος από τις εκλογές δηλαδή μέχρι το Φεβρουάριο. Και σχετικά με τις ημερομηνίες... Ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να αποφύγουμε ...ημερομηνίες που συμπίπτουν με θρησκευτικές ε, ή άλλες δημόσιες αργίες υπεύθυνοι ε, της Πεντηκοστής κλπ. Κάπου εκεί. Η διαδικασία τροποποίησης της ημερομηνία των εκλογών είναι ότι θα πρέπει να αποφασίσει το Συμβούλιο και να δώσει συγκατάθεση το Κοινοβούλιο. Θα έχουμε χρόνο λοιπόν να το σκεφτούμε. Αλλά είναι σημαντικό να τεθεί το θέμα της ημερομηνία. Διότι πρέπει να οργανωθούν οι εθνικές αρχές αντιστοίχως. Ίσως μπορεί να παρέμβει και ο Σάββατος Σέπλιν. Πολύ σύντομα σας παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μου κάνει εντύπωση η πρόταση του κυρίου Νταφ. Ιδίως για την ημερομηνία του Μαΐου. Έχει εμφανιστεί εκ νέου στην Επιτροπή μας αυτό το θέμα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό το θέμα και ούτε για το πρώτο σημείο έχω πρόβλημα. Το δεύτερο σημείο είναι καινούριο και εδώ βλέπω ένα σημαντικό πρόβλημα και δεν ξέρω, Άντριου, τι γνώμη έχεις εσύ. Νομίζω ότι μετατρέπει τη σχέση μεταξύ εκλογέων και μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί θα πρέπει κάποιο να πει ψηφίστε με, θα σα εκπροσωπώ στο Κοινοβούλιο ή ψηφίστε με γιατί μπορεί να γίνω επίτροπο. Αυτή η αβεβαιότητα νομίζω ότι αφαιρεί από τον σύνομο χαρακτήρα της διαδικασίας και στα μάτια των εκλογέων ε, δεν είναι σαφής η σχέση μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής και ο τύπος νομίζω, τα μέσα ενημέρωση νομίζω ότι θα το στυλιτεύσουν αξίζει να το συζητήσουμε, να το αναδιατυπώσουμε ίσως κάπως, να το εκφράσουμε διαφορετικά. Καταλαβαίνω ότι θέλεις να πεις ότι πρέπει να εκλέγονται τα μέλη της Επιτροπής, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι πρέπει να εκλέγονται μέσω του Κοινοβουλίου. Αυτό ε, το σημείο θέλω να συζητήσουμε. E cioè eh, a me abbastanza favorevolmente θα ήθελα να την κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, να πω ότι ε, γενικά ε, υπάρχει θετική αντιμετώπιση. Το να παίρνουμε δηλαδή το 50% της Επιτροπής από ε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει όμως να είναι κατάλληλοι για να γίνουν επίτροποι. Θα μπορούσε το Κοινοβούλιο να παρέχει, να προτείνει αυτούς τους μελλοντικούς επιτρόπους και θα επιλέγονται από τον πρόεδρο της Επιτροπής. Κάτι τέτοιο θα δούμε πώς μπορούμε να το διατυπώσουμε. Λοιπόν, στις 27 Νοεμβρίου που θα ξανασυνεδριάσουμε θα πρέπει να ε, ψηφίσουμε για το θέμα αυτό. Θα έχουμε και τις μεταφράσεις έτοιμες. Προτείνω λοιπόν 27 Νοεμβρίου το μεσημέρι ως προθεσμία κατάθεση των τροπολογιών για να είστε έτοιμοι για την ψηφοφορία. Θα το ξανασυζητήσουμε βέβαια το θέμα με τον Αντιπρόεδρο Σέρκοβιτ, γιατί θα είναι ένα από τα θέματα που θα αναφέρομαι στη συζήτησή μας. Να περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Πρώτα απ' όλα, ξεκινάμε με τις ρήτρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αμοιβαία άμυνα και αλληλεγγύη πολιτικές και επιχειρησιακές διαστάσεις. Ξεκινούμε λοιπόν. Ψηφίζουμε τα σημεία 4, 6, 12 και 16. Υπέρ. Διανατάσεως της χειρός παρακαλώ. Και κοντράριο. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 της κυρίας Γιαννάκου, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7, Σούλτς, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 έχει αποσυρθεί. Σημείο 7 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9 Γιάννης Μπαρνουέβο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβασμός α παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σημείο 8 του εισηγητού υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Τρασκόφσκι. Παρακαλώ ε, σηκώστε το χέρι σας υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Σημείο 9. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σημείο 10. Σημείο 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Σημείο 11 του εισηγητού. Σημείο 11 του εισηγητού. Υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται σημείο 13 υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 12 υπέρ. Προηγουμένως ο Πρόεδρος είχε πει τροπολογία 13 ενώ ήταν σημείο 13. Σημείο 13 λοιπόν τώρα είμαστε τροπολογία 12. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 να α, καταπίπτει. Το ίδιο και η τροπολογία 14 ή μήπως ε, η τροπολογία 14 δεν καταπίπτει, ρωτάει ο Πρόεδρος. Όχι, καταπίπτει. 14 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Και Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 Γιαννάκου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σημείο 15 του εισηγητού. Ε, μάλλον όχι. Το 16 εγκρίνεται, επομένως το σημείο 15 καταπίπτει. Τροπολογία 17, Γιάννιες Μπαρνουέβο, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18, υπέρ. Κατά. εγκρίνεται. Σημείο 17 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Σημείο 18 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Σημείο 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 που θα ψηφιστεί κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Αποχέ συγκρίνεται, 25 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται σημείο 20 του εισηγητού υπέρ κατά άποχες απόποχέ σημείο 1 του εισηγητού υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Σημείο 2. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 του συναδέλφου Σόλτς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 Ταρσκόφσκι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σημείο 3 κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 Γιάννης Μπαρνουέβο υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται τροπολογία 4 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται τροπολογία 5 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται σημείο 5 του εισηγητού υπέρ κατά Ε, πολύ κοντά ήταν το αποτέλεσμα, πάντως απερίφθη. Να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία της γνωμοδότησης, επί του συνόλου δηλαδή της γνωμοδότησης. Κατά. Κατά λοιπόν αποχές 14 υπέρ Αποχές, καμία αποχή. Εντάξει, εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Έκθεση Γκουαλτιέρη προς μια ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση. Να ξεκινήσουμε. Σημείο 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53 Hefner και θα ψηφίσουμε μονάχα την προσθήκη υπέρ. Έντεκα ψήφι υπέρ, κατά. 12 κατά, απερίφθη. Τροπολογία 55 υπέρ. Α, Κάτι ξεχάσαμε. Έχουμε την πρώτο, τον πρώτο συμβιβασμό. Έχουμε λοιπόν τον πρώτο συμβιβασμό του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ο συμβιβασμός. Δεν ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 55 ούτε το σημείο 31, ψηφίζουμε όμως την τροπολογία 54 αντάφ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται σημείο 32 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 56 νταφ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 58 κατά τμήματα ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Σημείο 33. Καταπίπτει. Έχει καταπέσει, δεν το ψηφίζουμε. Συμβιβασμός L. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα ψηφίσουμε το σημείο 34 το, τροπολογία 59, τροπολογία 60, τροπολογία 59, το σημείο 34 και την τροπολογία 60. Πηγαίνουμε απευθείας στο συμβιβασμό M υπέρ. Χωρίς μικρόφωνο, ο κύριος Γουαλτιέρη, χωρίς μικρόφωνο. Πρόεδρε, νομίζω ότι έγινε, μια έγινε ένα τεχνικό λάθος στην τροπολογία, μάλλον στη ψηφοφορία του 32. Ίσως δεν, δεν ήταν σωστές, σωστή η κατάλογη ψηφοφορίας ο συνάδελφος Δαρκόφσκι συμφωνεί να ξαναρχίσει η ψηφοφορία για το 32. Το κείμενο είναι απλό, αλλά όμως είναι πολύ σημαντικό για την έκθεση. Χωρίς μικρόφωνο Πρόεδρος. Ναι, ίσως εάν όλοι συμφωνούν να γυρίσουμε πίσω, εντάξει. Να το ξαναδούμε. Συμφωνείτε, συμφωνείτε να γυρίσουμε πίσω στην ψηφοφορία. Κύριε Ταρκόφσκι, συμφωνείτε να ξαναψηφίσουμε. Συμφωνούν όλοι να ξαναψηφίσουμε. Ε, Ο κύριος Νταφ. Μισό λεπτό παρακαλώ, λέει ο κύριος Νταφ. Εκτός μικροφώνου ο πρόεδρος. Μιλάω για το 32. Ναι, σημείο 32. Νταφ. Νταφ. Ε, η, έκβαση της ψήφου ήταν αρνητική. Τώρα ο Σνάφος Γκουαλτιέρη λέει ότι μάλλον δεν αναγνώστηκε σωστά το σημείο αυτό και ζητά επανάληψη του ψήφου, της ψηφοφορίας, συγγνώμη, ε, επανάληψη της ψηφοφορίας. Ο συνάδελφος Ταρκόφης συμφωνεί. Τι λέτε κύριε Ντάφη για το σημείο 32. Γραμματικό. Γραμματικό είναι το σφάλμα στα αγγλικά. Λέει privileges to proceed, ε, δηλαδή ότι, έχει, ε, ότι είναι κάτι σκόπιμο να γίνει. Αλλά τέλος πάντων γραμματικά αυτό είναι λάθος στα αγγλικά και γι' αυτό το λόγο λέει ο κ. Ε, φαντάζομαι ότι και το ΕΛΚΑ ήταν κατά. Και έχουμε την τροπολογία 57 ανταυτού. Εγώ έτσι το κατάλαβα. Εκτός μικροφώνου κάποιο σχόλιο. Όχι, όχι, όχι. Ε, αυτό ήταν διαφορετικό από το 57. Τζέραλτ, συμφωνείς. Λες τον κύριο Κούπερ. Ναι, ναι, εγκρίθηκε όμω το 57, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Εγκρίθηκε. Ναι, δεν νομίζω. Είναι ανώφελο να ξαναψηφίσουμε το 32 από τη στιγμή που εγκρίθηκε το 57. Ξαναέκλεισε το μικρόφωνο του Προέδρου. Χωρίς μικρόφωνο ο Πρόεδρος, δεν ακούν οι διερμηνείς. Α, Μα τι να κάνω, λέει ο πρόεδρο. Κλείνει το μικρόφωνο μου συνέχεια. Λοιπόν, συμβιβασμό M. Παρακαλώ, σηκώστε το χέρι σα όσοι συμφωνείτε. Συμβιβασμό M. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Καταπίπτουν λοιπόν οι τροπολογίε 61-62. Σημείο 35, τροπολογία 62, σημείο 35 και η τροπολογία 61 που είναι ταυτόσημη. Ψηφίσουμε λοιπόν το σημείο 36 υπέρ. Είναι ένα σημείο του συναδέλφου Τασκόφσκι. Κατά. βεσπίντο, Απερίφθη. Σημείο 37 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται με την ίδια πλειοψηφία. Τροπολογία 63 υπέρ. κατά αποχές Λοιπόν, να ξαναψηφίσουμε. Υπέρ. Υπέρ, υπέρ. Έντεκα ψήφοι υπέρ. Κατά. 12 ψήφοι κατά, επομένως απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία N λέει ο Πρόεδρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει ότι φτάνουμε στο σημείο 39 όλα τα ενδιάμεσα καταπίπτουν, καλύπτονται δηλαδή από το συμβιβασμό. Σημείο 39 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Σημείο 40. Έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 67. Ψηφίζουμε το 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 68. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός ο ψηφίζεται κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα χωρίς το η κοινωνική διάσταση. Μάλλον όχι. Κάνω λάθος λέει ο Πρόεδρος. Σε πάση περιπτώσει ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα που είναι μόνο ε, το, The Social Dimension υπέρ. Κατά. Έντεκα δώδεκα απερίφθη. 70, 41, 69 είναι στην, στο συμβιβασμό. Τροπολογία 71, DAF υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 72. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 73 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 74 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο παράρτημα. Τροπολογία 75 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 76 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 77 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 78 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 79 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Α, θέλετε επανάληψη της ψηφοφορίας επί της τροπολογίας 79. Πάρα πολύ ωραία. Τροπολογία 79 του κυρίου Ντάφα που ζητά διαγραφή. Υπέρ. Κατά. Ζητώ συγγνώμη, δεν είχαμε μετρήσει καλά ή δεν είχατε σηκώσει εσείς καλά τα χέρια σας, πάντως εγκρίνεται. Τροπολογία 79. Η 80 λοιπόν καταπίπτει και επομένως φτάνουμε στην τροπολογία 81, υπέρ. 81, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ναι, αλλά πρέπει να ψηφίζετε κανονικά, γιατί μερικές φορές δεν καταλαβαίνουμε τι θέλετε. Με ποιο τρόπο ψηφίζετε δηλαδή. Λοιπόν, τροπολογία 82 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι, απορρίπτεται. Πηγαίνουμε στο συμβιβασμό Α στον, ε, του εισηγητού υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Σημείο 1, τροπολογία 2 και η τροπολογία 1. Πρέπει να ψηφίσουμε μόνο το δεύτερο τμήμα που είναι συμβατό με το συμβιβασμό α υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σημείο 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε μαζί με την λέξη closer. Τροπολογία 3 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 λέει ο Πρόεδρος. Σημείο 3 έχουμε εμεί τον κατάλογο. Υπέρ. Κατά. να ψηφίζουμε γιατί αλλιώς δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός B. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σημείο 4. Τροπολογία 5. Αυτά είναι μέσα στο συμβιβασμό. Ε, φτάνουμε στο συμβασμό C δύο τμήματα. Πρώτα ψηφίζουμε χωρίς το The Social Dimension, όπως και την προηγούμενη φορά λοιπόν. Ψηφίζουμε το σύνολο πλην της κοινωνικής διαστάσεως. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερη ψηφοφορία μόνο τα The Social Dimension. Υπέρ. κατά, κατά, δώδεκα προς 11 απορρίπτεται. Τροπολογία 6, σημείο 5, τροπολογία 7 καλύπτονται από το συμβιβασμό. Σημείο 6 υπέρ. Σημείο 6 υπέρ. κατά χες νομίζω πως εγκρίνεται ναι, εγκρίνεται κύριε πρόεδρε ίσως μέτρησα εγώ άσχημα αλλά στον συμβιβασμό uh, εγώ μέτρησα ανάποδα από το δικό σας αποτέλεσμα μπορείτε στο δεύτερο τμήμα ναι, the social dimension μπορείτε να επαναλάβετε την ψηφοφορία παρακαλώ χωρίς μικρόφωνο ο πρόεδρος Νομίζω ότι με μεγάλη φροντίδα μετρήσαμε τις ψήφους. Ναι, αλλά αυτό αρχικά ήταν τροπολογία, ενώ τώρα μπήκε στο κανονικό κείμενο και επομένω σε μερικού καταλόγου ψηφοφορία έχει το αρνητικό πρόσημο, ενώ θα έπρεπε τελικά να είχε μπει το θετικό. Ίσως, ίσως κάποιοι δεν μην το κατάλαβαν καλά και ίσως γιατί ο συνάδελφος ζητάει να, να ξαναψηφίσουμε στο δεύτερο τμήμα. Λοιπόν, ζητάτε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία στο δεύτερο τμήμα, δηλαδή ε, αυτή την ψηφοφορία που αφορά το The Social Dimension. που αφορά το συμβιβασμό C. Ε, αν έχετε αμφιβολία σας επαναλάβουμε. Εντάξει. Ψηφίζουμε λοιπόν για να επιβεβαιώσουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, συμβιβασμός C, το δεύτερο τμήμα, δηλαδή μόνο το, η, τις λέξεις the social dimension. Κατά. Δώδεκα κατά. Καλά είχαμε μετρήσει. Επομένως επιβεβαιώνεται η αρνητική έκβαση. Τροπολογία 8. Τροπολογία 8. Χωρίς μικρόφωνο, ο κύριος Γκουαλτιέρη, δεν ακούμε δυστυχώς. Έντεκα υπέρ, δώδεκα κατά. Δώδεκα. Comunque le ho contate anch'io le mani alzate, non è che... Eh. Vabbè, allora siamo all'emendamento 8. Λοιπόν, τροπολογία 8, υπέρ. Υπέρ. Τροπολογία 8. Ε, τροπολογία Χέφνερ. Che fa il PPE? Immediatamente 8, non si capisce. Votano 5 del PPE. Ecco, voto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vabbè, è approvato. Εγκρίνεται. Ε, σημείο 7. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Chi è contrario? Ε, τροπολογία 12. 12 ε, κατά, άρα απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Ε, συγγνώμη του κυρίου Νταφ, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ. <clears throat> Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Σημείο 8 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 16 υπέρ δώδεκα υπέρ κατά Εγκρίνεται. Σημείο 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Ε, ψηφίζουμε, το ψηφίζουμε ως προσθήκη υπέρ αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός D του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. τροπολογία 19, σημείο 10, τροπολογία 20 καλύπτονται. Πρέπει να ψηφίσουμε όμως το σημείο 11 υπέρ. Σημείο 11 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21 να κάνουμε μία επαλήθευση. Μία επαλήθευση για το σημείο 11. Ωραία, σημείο 11 λοιπόν. Σημείο 11 υπέρ. Κατά. Eh, Απερίφθη λοιπόν. Τροπολογία 21 του Χέφνερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12, σημείο 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός ή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πάμε απευθείας στο σημείο 14. Όλα τα προηγούμενα καταπίπτουν. Καλύπτονται δηλαδή. Σημείο 13, τροπολογία 22, τροπολογία 23, σημείο 13. Λοιπόν, να ψηφίσουμε πρώτα για, το, για το, την τροπολογία 24 Χέφνερ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός F. Επειδή είδα ότι... Ναι, είναι σημείο 15, το πέρασα λίγο, γιατί βλέπω ότι αργούμε, τέλος πάντων. Σημείο 15 υπέρ, κατά, απερίφθη. Συμβιβασμός F υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και επομένως θα περάσουμε το σημείο 16, την τροπολογία 26 και την τροπολογία 27 και θα φτάσουμε απευθείας στην τροπολογία 28 του εισηγητού υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Νταφ υπέρ. Κατά. Όχι. Να μετρήσουμε πρώτα. Κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. Χωρίς μικρόφωνο κύριο Νταφ. να επαληθεύσουμε, ναι, ωραία, να ξανακάνουμε την ψηφοφορία. Τροπολογία 29 DAF υπέρ. Κατά. 11 υπέρ, 12 κατά, επομένως απορρίπτεται. Τροπολογία 30 DAF υπέρ. κατά Απερίφθη λοιπόν. Τροπολογία 31 ντάφι πέρ Κατά. Ίδια πλειοψηφία. Και απορρίπτεται. Σημείο 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σημείο 18, εδώ έχουμε και κάποιο κάτι άλλο με προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά 32. δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σημείο 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σημείο 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 34 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 35 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Δεν κατάλαβα. Τροπολογία 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σημείο 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 36 υπέρ. κατά απόχες εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, Συμβιβασμό H λέει ο Πρόεδρος, αλλά μάλλον βιάζομαι λέει, βιάζομαι ναι. Έχουμε πρώτα το σημείο 22 του εισηγητού, υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Τώρα έχουμε το συμβιβασμό H, υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. Και πάμε απευθείας Πάμε στο σημείο 24 του εισηγητού. Υπέρ. Κατά. Έντεκα προς έντεκα. Αλλά να το ξαναδούμε. Σημείο 24. Ξανά. Υπέρ. Κατά. Επομένω απορρίπτεται. Με 12 ψήφου κατά τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ. Κοντράρι. Κατά. Αποχές. è approvato. Εγκρίνεται λοιπόν. Ναι, εγκρίνεται. Σημείο 25 του εισηγήτου υπέρ. Contrari. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 41. Υπέρ. Νομίζω ότι το 41 πρέπει να ψηφιστεί. Το 41 ή το 42 λέει ο πρόεδρος. Το 41. Ναι, το 41, το 41. Νομίζω ότι είπα 41. Λοιπόν, υπέρ του 41. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται Μα, ε, λέει ο πρόεδρος εγκρίνεται συγγνώμη εγκρίνεται συμβιβασμός π παρακαλώ το χέρι σας να σηκώνετε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σημείο 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σημείο 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σημείο 28 υπέρ. Κατά. Έντεκα προς 12 απορρίπτεται. Σημείο 29 υπέρ. Η ίδια πλειοψηφία από ό,τι βλέπω. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 50. Υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 51 κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε τώρα την τελική ψηφοφορία επί της γνωμοδοτήσεως. Για να δούμε. Κατά. Δεκαοκτώ υπέρ, οι υπόλοιποι κατά, αποχές. Α, για να δούμε πώς είναι και η κατά, λέει ο πρόεδρος. Κατά. Τρεις ψήφοι κατά. Αποχές καμία. Ολοκληρώσαμε και την ψηφοφορία αυτή. Συγχαρητήρια γιατί όλοι δουλέψαμε μεν λέει ο Πρόεδρος αλλά ο, και ο κύριος Κουελτιέρη περισσότερο από όλους. Ναι, προηγουμένως στην τελική ψηφοφορία δεν καταγράψαμε την αποχή του κυρίου Σόλτς.

Να, ψηφίσουμε τώρα, να συνεχίσουμε. Ενδιάμεση έκθεση. σχετικά με το πολιετές δημοσιονομικό ε, πλαίσιο. Είναι η γνωμοδότηση του κ. Ταρκόφσκη. Γρήγορα όμως πρέπει να πάμε. Τροπολογία 4. Κατά. Να ψηφίσουμε, συνάδελφε Γκουαλτιέρη. Να ψηφίσουμε. Τι ψηφίζουμε. Α, την έκθεση Ταρκόφση σχετικά με την ενδιάμεση έκθεση εν της ε, ε, διαδικασίας έκβασης, της, ε, ε έγκρισης του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 4 υπέρ κατά. Εγκρίνεται. Ναι. Τροπολογία 5 υπέρ κατά πρέπει να μετρήσουμε. Κατά. Μάλλον όχι, να ξαναρχίσουμε λέει ο πρόεδρος, γιατί είμαστε λίγο κουρασμένοι φαίνεται και αφαιρεθήκαμε. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός Α. Τι έκανα. Α, ξεχάστηκα. Βλέπω αυτό το μεγάλο πλαίσιο που αφορά τη συμβεβαστική τροπολογία και το μάτι μου δεν πιάνει την άλλη, το μικρό τετραγωνάκι. Λοιπόν, ε, τροπολογία 9 της παραγράφου 24 υπέρ. Κατά. Πρέπει να μετρήσουμε, πρέπει να μετρήσουμε λέει ο Πρόεδρος. Άρα, Adesso il compromesso A, favorevoli. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι 10, οι 11 έχουν καλυφθεί. Η τροπολογία 12, 12 υπέρ. Κατά. 11 υπέρ, 11 κατά. Δεν εγκρίνεται επομένως. Θα επαναλάβουμε, θέλετε να επαναλάβουμε. Ήταν σαφής η ψηφοφορία ή όχι. Κύριε Πρόεδρε, να διευκρινίσουμε ε, κάποια σημεία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ. Γιατί νομίζω ότι αρκετές ψηφοφορίες μοιάζουν να είναι πολύ αμφίσιμες. Θα ήταν πιο απλό να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Όπως θέλετε. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, όχι, όχι. 11 ή 12 λέει ο Πρόεδρος. 12, 12 ψηφίζουμε. Τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 12. Εψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Λοιπόν, εψήφισαν 21 βουλευτές, 9 ψήφοι υπέρ, 12 κατά, επομένως απερίφθη. Περνάμε στην τροπολογία 13. Θέλετε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Θα Επειδή δεν τα βλέπουμε, δεν τα διαβάζει. Πρόεδρος, θέλετε να συνεχίσουμε με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ό,τι θέλετε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 13. Τροπολογία 13 δεν ψηφίζουμε, λέει ο πρόεδρο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Αποτέλεσμα. Εννέα ψήφοι υπέρ, 12 κατά, απορρίπτεται και μία αποχή. Ψηφίζουμε την τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. 15. Τροπολογία 15, ναι. ναι. Άρχεται η ψηφοφορία. È Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. È chiusa la votazione. È Απερίφθη. Ψηφίζουμε την τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Λοιπόν, να ψηφίσουμε την τροπολογία 17. Εγώ νόμιζα ότι αυτό ψηφίσαμε, λέει ο πρόεδρος, μάλλον μπερδεύτηκα. Λοιπόν, τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεν εγκρίνεται. Είναι 11 ψήφοι υπέρ, 11 ψήφοι κατά. Επομένως <coughs> απορρίπτεται. <coughs> Τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία 19 ψήφοι υπέρ 3 ψήφοι κατά. Ψηφίζουμε την τροπολογία 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Τώρα λοιπόν κυρίσω το πέρας της ψηφοφορίας. Δεν εγκρίνεται. Πάλι 11 ψήφοι υπέρ, 11 κατά, επομένως ε, δεν εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τρεις ψήφοι υπέρ, 18 κατά μία αποχή. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Συγγνώμη, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Εγκρίνεται. 20 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά. Αυτή ποια τροπολογία ήταν πάλι που ψηφίζαμε. Η τροπολογία 1. Πάρα πολύ ωραία. Τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Δεν εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 18 ε, ψήφοι υπέρ, 3 ψήφοι κατά, μία αποχή. Θε, ε, κώδικας διοικητικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, να προχωρήσουμε με την διατάσταση του και βλέπουμε. Κώδικας διοικητική διαδικασία είναι γνωμοδότηση της κυρίας Γέτερ Μάκη. Τροπολογία 14 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 μέσα Σμιτ υπέρ. Κατά. 11 υπέρ 12 κατά, εντάξει. 12 ε, υπέρ 11 κατά, εγκρίνεται μάλλον. Όχι, θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση. Τροπολογία 15 Μέρσερ Σμιτ, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, πονιάμε votazione per Ψηφίζουμε την τροπολογία 16. Ανατάσσεως της χειρός η ψηφοφορία. Θέλετε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μα δεν είπαμε πρώτα διανατάσσεως της χειρός. Εάν θέλετε ηλεκτρονική ψηφοφορία, κανένα πρόβλημα. Αλλά είναι πιο αργός, ε, αργός τρόπος η ηλεκτρονική ψηφοφορία. E chiusa la Πέρα ε, approvato. Εγκρίνεται. Emendamento 17. 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Πού είναι το 17. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Εγώ επιμένω, λέει ο Πρόεδρος, ότι πρέπει πρώτα να κάνουμε ε, διανατάσεις της χειρός. Θέλετε να δοκιμάσουμε διανατάσεις της χειρός. Τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Μα είπα ε, ηλεκτρονική τελικά. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 19 Ράντζελ. Πέρας. Δεν εγκρίνεται 10 ψήφοι υπέρ, 10 κατά. Η ισοψηφία επομένως δεν εγκρίνεται. Τροπολογία 20 Ραντζέλ έρχεται η ψηφοφορία. Eh, non abbiamo il segnale. Εγκρίνεται. Λέω πρώτος, έχω την, την ε, ψηφορία 21. Ράντζελ. Ψηφίζουμε. Πέρα. Εγκρίνεται. 22. Ράντζελ. Ψηφίζουμε. Πέρα. Εγκρίνεται. 23. Γκουαλτιέρι. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 24. Γιαννάκο. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 25. Ραντζέλ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτωται. 10-10. 26. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην τροπολογία Παραθμανένα για τι αιτιολογικές παραγράφους. Γκουαλτιέρη. Δύο-δύο ψηφορίες θα κάνουμε. Ε, κατά διαίρεση, πρώτα-πρώτα, γιατί για το πρώτο κομμάτι σηκώστε το χέρι. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ποιοι είναι υπέρ για το δεύτερο τμήμα, σηκώστε το χέρι. Αποχές, κατά, εγκρίνεται. Δύο. Γκουαλτιέρη. Ποιο είναι υπέρ, σηκώ στο το χέρι, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρία, μέσο Σμιτ. Σηκώστε το χέρι υπέρ. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Ψηφίζουμε. Πέρα. Εγκρίνεται. Συμβαστική Α Υπέρ. Σηκώστε το χέρι. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, έξι. Μέσο σμιτ. Σηκώστε το χέρι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έπτα. Ραντζέλ. Ποιοι είναι υπέρ, Σηκώστε το χέρι. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Περ, σηκώστε το χέρι, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 έχει καλυφθεί ήδη, επομένως δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε. Τροπολογία 9 επίσης. Τροπολογία 10 Γκουαλτιέρη, παρακαλώ, σηκώστε το χέρι σας. θέλετε ηλεκτρονική ψηφοφορία, εντάξει. Πέρα της ψηφοφορίας Απερίφθη. Τροπολογία 11 Γκουαλτιέρη υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12 Γκουαλτιέρη υπέρ, σηκώστε το χέρι σας όσοι είστε υπέρ, κατά, κα, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13 Γκουαλτιέρη υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία διολεκτρονικής ε, ψηφοφορίας. Άρχεται η ψηφοφορία για την τελική ε, ψηφοφορία λοιπόν. Εψήφισαν όλοι. Για να δούμε το αποτέλεσμα. Οι 22 υπέρ, καμία, ψήφος κατά, καμία αποχή. Πολύ ωραία. Να συγχαρούμε την κυρία Γέτεν Μάκη. Έχουμε τώρα το σημείο 15 θέσμιση του προγράμματο Ευρώπη για του πολίτε για την περίοδο 2014-2020. Μα πόσε τροπολογίε έχουμε, πόσε ψηφοφορίε ψηφοφορίες έχουμε, λέει ο Πρόεδρος. Πολλές. Ce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 ψηφίζοντας ε, επί της ε, εκθέσεως Hefner Ευρώπη για τους πολίτες 2014-2020. Να ξεκινήσουμε διανατάσεως της χειρός τροπολογία 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 του εισηγητού πάντα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κύριε Πρόεδρε, μήπως μπορούμε να ψηφίσουμε αμπλόκ όλη τη σειρά. Αυτό είχα ζητήσει και εγώ, αλλά το ΕΛΚ δεν το δέχτηκε. Δηλαδή να ψηφίσουμε μέχρι να υπάρχει αμφιλεγόμενη ψήφος. Ε, φαίνεται ότι στο πρώτο μπλοκ των τροπολογιών δεν υπάρχει αντίθεση. Όχι. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα, λέει ο Προεδρο. τι θέλετε. Θέλετε πάντω ηλεκτρονική ψηφοφορία για το 16. Τι, ε, ζητάτε ηλεκτρονική ψηφοφορία, λέει ο προεδρο Όχι. Να, να συνεχίσουμε λοιπόν διανατάσσεω τη χειρός. Τροπολογία 16 υπέρ. <coughs>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 ένα της κυρίας Γιαννάκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της ε, τροπολογίας 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ. Ξεχάστηκε, συνάδελφε Γκουελτιέρη. Εγκρίνεται.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 κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 Τελική ψηφοφορία επί του συνόλου της ε, εκθέσεως. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, εντάξει, ναι, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 19 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Γιάτερ Μέκη. Α, ναι, μπερδεύτηκα, λέει ο πρόεδρος. Δεν ήταν έκθεση της κυρίας Γιατερμάκη. Ήτανε του κυρίου Χέφνερ, που κι αυτός δεν λέγεται Χάφνερ, λέγεται Χέφνερ, οπότε δεν πειράζει. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία.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 Θέλετε να, βάλουμε, να ψηφίσουμε πρώτα το, το τελικό για το σχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με την ε, τσεχική δημοκρατία του κυρίου Νταφ. Εντάξει, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Απερίφθη. 10 υπέρ, 12 κατά. Είναι πολύ ευχαριστημένος ο κύριος Νταφ να μας δώσετε και τα αποτελέσματα. 10 ψήφοι υπέρ, 12 ψήφοι κατά, μία αποχή. 10 ψήφοι υπέρ, 12 κατά, μία αποχή. <laughs> Συγχαρητήρια στον εισηγητή λοιπόν. Ναι, ναι, συγχαρητήρια στον εισηγητή, άψογα, πάρα πολύ ωραία. Allora, fare Έχουμε την τελευταία έκθεση. Ευτυχώ που τελειώνουμε λίγο πρόεδρο γιατί τα μπέρδεψα λίγο σήμερα τροποποίηση του άρθρου 181 κτλ. κτλ του συναδέλφου Ήλτσεφ. Νομίζω ότι καλύτερα είναι να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν ψηφοφορία, να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Συμβιβαστική τροπολογία Α. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν είναι εδώ το ΕΛΚ. Απουσιάζει πλήρως. Συμβιβαστική τροπολογία Α. Πέρα τη la Πέρας της Απερίφθη πανηγυρικά. πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 8 γιατί δεν έγινε δεχτή η συμβιβαστική τροπολογία. 8 λοιπόν υπέρ. Η υπέρ της τροπολογίας 8. Κατά. Απερίφθη. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Υπέρ. Τροπολογία 1. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 του εισηγητού. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 και τροπολογία 9. Είναι ταυτόσιμες τροπολογίες αυτές. Υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Υπέρ της τροπολογίας 3. Κατά. Απερίφθη. Όχι, εγκρίνεται, λέει ο πρόεδρος, διορθώνει. Εγκρίνεται, εγκρίνεται η τροπολογία 3 του εισηγητή. Τροπολογία 4 του εισηγητού. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός B. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και επομένως καταπίπτουν ή ενσωματώνονται οι τροπολογίες 11 και 5. Συμβιβαστική τροπολογία C. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 12 λοιπόν έχει καταπέσει και η τροπολογία 6 και η τροπολογία 13. Επομένως ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία, η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τελική μας ε, ψήφο πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 19 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά, δύο μονάχα αποχές. Συγχαρητήρια, κύριε Σνάλφε Ήλτσεν. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η διαδικασία της ψηφοφορίας. Πρόεδρος, μπορούμε να ξαναρχίσουμε λοιπόν τις εργασίες μας. Παρακαλώ πολύ, θέλω να σας ζητήσω να καθίσετε, να συνεχίσουμε τις εργασίες της Επιτροπής μας. Και όσοι θέλουν να κάνουν ψηλοκουβέντα, παρακαλώ πολύ να την κάνουν εκτός της αιθούσης. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, Αντιπρόεδρο, ε, κύριο ε, Μάρο Σεύκοβιτς και να τον να του ζητήσω συγγνώμη και εξ ε, του εποφαινομένου αλλά και εξ ονόματος όλων σας ε, για την ε, καθυστέρηση με την οποία τον υποδεχτήκαμε. Θα ήθελα να πω ότι το θέμα των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και η χρηματοδότησή τους είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για τη δική μας Επιτροπή. Μετά από πολλές συζητήσεις για το θέμα αυτό θεωρούμε ότι αυτά τα ζητήματα είναι απολύτως συνδεδεμένα με την προώθηση της Ευρώπης. Ε, ήδη είχαμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει θέση και στην προηγούμενη ε, θητεία βάσει προτάσεως του συναδέλφου Γιολάινεν. Και τώρα έχουμε την πρόταση της κυρίας Γιαννάκου θα ήθελα να σας υπογραμμίσω λοιπόν την σημασία την οποία να αποδίδουμε στο θέμα αυτό ε, και θα δώσω αμέσως το λόγο στον ε, Επίτροπο Σεύκοβιτς ε, εκφράζοντας βεβαίως και την λύπη μου διότι δεν θα έχουμε στη διάθεσή μας όλο τον χρόνο που είχαμε προβλέψει. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Από τη βλέπω είχατε πολλή δουλειά σήμερα το πρωί και είχατε και μακράς ψηφοφορίες αλλά να η ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτήν την τόσο παραγωγική, δημιουργική, χρήσιμη συζήτηση. Το θέμα αυτό είναι σημαντικό για όλους μας και σας παραπέμπω στην ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και στη συζήτηση που ακολούθησε, διότι τότε ε, ξεκάθαρα προέκυψε το τι χρειαζόμαστε στο μέλλον, να αντιμετωπίσουμε την κρίση, να έχουμε περισσότερη πολιτική νομιμοποίηση στην Ευρώπη, γιατί σίγουρα ε, χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη για τους ε, Ευρωπαίους. Νομιμοποίηση επομένω πολιτική. Και προς τούτο θα πρέπει να εξελίξουμε τα θεσμικά όργανα, να βελτιώσουμε τη λειτουργία της Ένωσης και έτσι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις σημερινές και αυριανές προκλήσεις. Θα θυμάστε επίσης ότι ήταν ξεκάθαρο το ότι τα πολιτικά κόμματα επιβάλλεται να γεφυρώσουν αυτό το κενό που δημιουργηθεί μεταξύ της εθνικής πολιτικής και της ευρωπαϊκής πολιτικής και ότι θα πρέπει επίσης κάτι να γίνει όσον αφορά την ικανότητα της Ένωσης να αναλαμβάνει δράση. Έχουμε κάποιες προτάσεις για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ιδρύματα. Οπότε είπαμε ότι έχουμε κάποιο πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να ολοποιήσουμε αυτές τις φιλοδοξίες μας. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Γιαννάκο η οποία διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο σε σχέση με το θέμα τούτο, σε σχέση με την διεκπαιρέωση, την υλοποίηση των όσων είχαμε ως ιδέες και επίσης όπως είπε και ο πρόεδρος και είχαμε πει και πριν τις διακοπές ότι προσπαθήσαμε να καλύψουμε τις προτάσεις μας, τις δικές σας προτάσεις, τις δικές σας ιδέες και αυτά τα οποία είχε πει ε, στο έγγραφο της 20 Απριλίου η κυρία Γιαννάκου. Επίσης, έχουμε συγκεκριμένες ε, λύσεις να προτείνουμε κατόπιν του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου επί της εκθέσεως Γιαννάκου. Έτσι θα προχωρήσουμε και έχουμε αυτές μας προτάσεις για ε, τον σεβασμό των ε, αξιών της Ευρώπης, όπως λέμε την δημιουργία ε, ενό πλαισίου σύμφωνα με το οποίο τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα έχουν προσβασιμότητα στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ναι, εδώ με τώρα, έχουμε μια ολόκληρη δεσμή προτάσεων να κατεβάσουμε και σας εξηγώ. Έχουμε ναι, να προτείνουμε έναν κανονισμό. Με τον οργανισμό αυτό θα θεσπιστεί ε, κάποιο είδου καταστατικό ευρωπαϊκό που θα διέπει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και επίσης τα σχετικά πολιτικά ιδρύματα. Μια νέα επομένω ευρωπαϊκή νομική προσωπικότητα η οποία θα είναι αναγνωρισμένη σε όλα τα κράτη-μέλη. Κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι καινοτομία. Και θα αναγνωρίζονται κόμματα και ιδρύματα τα οποία θα πληρούν κάποιε προποθέσει, κάποια πρότυπα και κυρίω να ενασέμονται τι αξίε που είναι τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, σεβασμό της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας, δημοκρατία, ελευθερία, ισότητα, κράτος δικαίου και σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και βέβαια, δεν θα πρέπει να έχουν και οδοσκοπικό σκοπό. Παραγνωρίζεται επομένω μόνο κόμματα και ιδρύματα τα οποία θα διέπονται από κανόνε διαφάνεια, εσωτερική λειτουργία του κόμματο και δημοκρατική επιλογή των υποψηφίων ε, αυτών που κατέχουν διάφορες διοικητικές θέσεις κλπ. Και θα πρέπει επίσης τα κόμματα αυτά να σέβονται τις, είπαμε, τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες και αυτό θα ενδυναμώσει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα μπορεί το Ευρωπαϊκό να αναλαμβάνει δράσει σχετικώ. Τώρα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση αυτών των κομμάτων και ιδρυμάτων. Προτείνουμε κάποιες μεταβολές σε δύο επίπεδα. Πρώτα-πρώτα, με αυτό το καταστατικό θα έχουμε επίσης και ένα ολόκληρο πλαίσιο, ολοκληρωμένο για τη χρηματοδότηση, για τις δαπάνες, τις συνδρομές, τις δωρεές σε σχέση με τα κόμματα. Περισσότερη διαφάνεια, και καθώς θα και κάποιες κυρώσεις. Επίσης θα έχουμε, θέλουμε περισσότερη ευελιξία όσον αφορά αυτή τη χρηματοδότηση και θα ανέβει, το κατόφλι ε, σε σχέση με τα 25.000 ευρώ και το κατόφλι για τις δωρεές. Ε, επίσης, σύμφωνα με το όριο αυτό, θα ορίζεται ποιες δωρεές θα, πρέπει να, μπορούν να μείνουν ανώνυμες επίσης. Θέλουμε να αλλάξει το ισχύον σύστημα του χρηματοδοτικού κανονισμού και θα έχουμε ένα νέο κανονισμό. Θα υπάρχει διαφορετικό κεφάλαιο, ειδικά που θα διέπει τα κόμματα ε, και θα ρυθμίζει τα των ε, ιδιοτύπων αυτών συνδρομών προς τα κόμματα. Θα έχουμε αυτό το σχέδιο κανονισμού επομένω και αυτό το σχέδιο θα γίνει νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής μόλις αρχίσει να ισχύει από τους συνομοθέτες ο νέο δημοσιονομικός κανονισμός το οποίο ελπίζω ότι θα συμβεί κάποια στιγμή περί τα τέλη του μήνα. Έτσι θα έχουμε τέτοιο τέτοια, τέτοια καταστροφικό που θα διέπει τα κόμματα, θα λέει για τους ιδίους πόρους των κομμάτων, θα λέει για το κατά πόσον ε, θα μπορούν να κάνουν μεταφορά των ε, εισφορών της Ένωσης μέχρι δύο χρόνια. Θέλουμε να υπάρχουν όσο γίνεται περισσότερα δικαιώματα συγχρηματοδότηση από τον ε, προπολογισμό και επίση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να υπάρχει το, το, η λεγόμενη προπόθεση του να έχει το κόμμα έναν ευρωβουλευτή για να μπορεί να έχει πρόσβαση στη Ε, χρηματοδότηση. Και είπαμε ότι για μα είναι αυτό σωστό κριτήριο με δεδομένη τη συνθήκη που αναγνωρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν το κομβικό σημείο έκφραση των Ευρωπαίων. Τώρα. Για να δούμε τώρα που θα στρέψουμε την προσοχή μας, αλλά και τις προσπαθειές μας. Σε σχέση δηλαδή με την ταχεία έγκριση της δέσμης των προτάσεων. Εμείς εδώ έχουμε κάποιους φιλόδοξους στόχους. Σε σχέση με τη θέση σε ισχύ αυτού του νέου κανονισμού. Και θέλουμε να εγκριθεί, να τεθεί σε ισχύ από 1η Σεβδόμου 2013. Νομίζω ότι αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο θέλουμε, πόσο πιστεύουμε σε αυτό το νέο πλαίσιο. Και βεβαίως και εσείς θέλετε πριν τις ευρωεκλογέ να λειτουργεί αυτό το πλαίσιο τις εκλογέ του 2014 δηλαδή. Ήδη έχω διαβάσει το χρονοδιαγραμμά σας, θέλετε δηλαδή τον Ιανουάριο να συζητήσετε το κείμενο αυτό στην Επιτροπή και μετά τον ε, τριμερή διάλογο, Μάρτιο-Απρίλιο, θέλετε να έχει υποβληθεί το κείμενο στην ε, Ολομέλεια. Πάρα πολύ φιλόδοξο σχέδιο και νομίζω ότι μα βρίσκει σύμφωνο. Ήδη έχουν αρχίσει οι επαφέ, οι συζητήσει με τα κράτη-μέλη. Υπέβαλα τι προτάσει μα στου ε, Υπουργού Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων πριν από λίγε εβδομάδε υπό Κυπριακή Προεδρία. Τα είπαμε στο σχετικό συμβούλιο η Προεδρία συμφωνεί ότι θα προχωρήσει ταχαίω για τα θέματα αυτά. όπω είχε υποσχεθεί στην, στο Συμβούλιο Γενικών Προθέσεων και στην ομάδα εργασία, η οποία έχει συνέλθει τρει φορέ ήδη και την και τέταρτη αυτή τη βδομάδα, όπω προβλέπετε, όλα αυτά επομένως ε, για να ζητηθούν αυτά τα ζητήματα με στόχο την, ε, μάλλον τη βάση τη απόφαση του 27 Σεπτεμβρίου. Αυτά όσον αφορά τις προτάσεις, αυτά όσον αφορά τη θέλησή μας να προχωρήσουμε ταχαίως και έτσι να έχει κλειστεί το θέμα τον, το, το, το, καλοκαίρι του χρόνου. Πάντως κάποια κρατημέλη επικρίνουν τις προτάσεις μας ιδίω όσον αφορά τα μέτρα ευελιξίας για την χρηματοδότηση από τον προπολογισμό. Γι' αυτό και θα ήθελα να προτείνω στην Επιτροπή σας ε, και στους εισηγητές να έρθουν σε επαφή, να αρχίσει διάλογο συντατικά με, με προς πάσα κατεύθυνση και κυρίως προς τα κράτη-μέλη ε, ε, και αυτή η συζήτηση πιστεύω θα είναι πάρα πολύ θετική για το θέμα μας διότι νομίζω ότι έχετε πάρα πολύ βάσιμα επιχειρήματα ούτως ώστε να διασκεδάσετε κάθε αμφιβολία και κάθε παρεξήγηση να την άρετε και εγώ και οι υπηρεσίε της Κομισιόν γενικότερα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευκολύνουμε την διαδρομή σας και να υπάρξει ταχεία επομένως ε, συμφωνία όσον αφορά αυτές τις προτάσεις. Πιστεύουμε κράτοντα ότι είναι πολύ σημαντικέ αυτέ οι προτάσεις και άλλωστε η συντριπτική μας πλειοψηφία στην Επιτροπή ενέκρινε αυτές τις προτάσεις. Άρα θέλουμε να έχει ολοκληρωθεί προσπάθειά μας μέχρι τον Ιούλιο του 2013 και να υπάρχει μετά το περιθώριο των χρονικών, να το χρησιμοποιήσουν αυτό το καινούριο πλαίσιο τα ευρωπαϊκά κόμματα πριν τις ευρωεκλογές του 2014. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ λέει ο για τα όσα μας είπατε. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους αλλά θα πρέπει να δώσουμε το λόγο βέβαια και στην κυρία Γιαννάκου, η οποία έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο σε αυτή την θητεία και επίση τον συνάδελφο Γκερέρο, ο οποίος ε, είναι ο εισήγητή όσον αφορά τον χρηματοδοτικό κανονισμό. Και κατόπιν θέλαμε το λόγο οι άλλοι συνάδελφοι. Ε, κυρία Γιαννάκο, αν θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κύριο Σεύκοβιτς γιατί ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Κοινοβουλίου με τον καλύτερο τρόπο προετοιμάζοντας την έννοια του καθεστώτος του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος. κύριε Επίτροπε, ε, ειλικρινά σας ευχαριστώ και ευελπιστώ στη συνεργασία σας μέχρι τέλους. Ε, θέλω να σχολιάσω το εξής. Στα κράτη-μέλη είναι πολύ γνωστός ο όρος Ευρωπαϊκό Κόμμα στα έντυπα, στην τηλεόραση παντού ακούγεται το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό Κόμμα της Αριστεράς, των Φιλελευθέρων κτλ. Υποθέτω ότι οι πολίτες φαντάζονται πως τα κόμματα αυτά έχουν ένα συγκεκριμένο καθεστώς κόμματος. Εάν μάθουν ότι τα κόμματα αυτά είναι περίπου διεθνείς μη κυβερνητικέ οργανώσεις στο Βέλγιο, ομολογώ ότι θα εκπλαγούν δυσάρεστα. Έτσι λοιπόν αυτή την ώρα προσπαθούμε να κάνουμε κάτι που έπρεπε να έχει ήδη γίνει για να συμπληρώσει την αξία και το συμβολισμό που πρέπει να έχει ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και μάλιστα σημειώνοντας ότι η Επιτροπή μας έχει δεχθεί ότι τα κόμματα αυτά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δέχονται ακόμα και απλά μέλη ως μέλη τους. Απ' την άλλη πλευρά μας χρειάζεται ένα νομικό καθεστώς, sui generis θα έλεγα, το οποίο να μπορεί μέσω του κανονισμού να δίνει νομική προσωπικότητα στα κόμματα σε όλα τα κράτη-μέλη και φυσικά και τη δυνατότητα αν ένα κόμμα θέλει να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος να το κάνει. Επομένως η συζήτηση με το Συμβούλιο που ανέφερε ο κύριος Επίτροπος ασφαλώς είναι αναγκαία. Θέλω να σημειώσω κύριε Πρόεδρε ότι εδώ είχαμε πει ότι τα κόμματα δεν ζητούν περισσότερα χρήματα. Ζητούν ένα πραγματικό νομικό καθεστώς που δεν θα τους φέρνει σε αντίθεση με την ομοθεσία των κρατών μελών και θα τους δίνει την νομική προσωπικότητα που χρειάζεται ώστε να φαίνεται ότι και οι πράξει τους σε όλα τα επίπεδα είναι διαφανείς. Επομένως τα κράτη-μέλη που ανησυχούν και αντιλαμβάνομαι ποια κράτη-μέλη ανησυχούν και νομίζουν ότι αυτός ο κανονισμός γίνεται για να πάρουν τα κόμματα περισσότερα χρήματα Νομίζω ότι κάνουν λάθος. Η προσπάθειά μας έχει θεσμικό χαρακτήρα. Και αυτό επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, ξέρω ότι και ο συνάδελφος Γκερέρο συμμερίζεται αυτές τις απόψεις. Είναι κυρίως το θεσμικό κομμάτι που θέλουμε να ικανοποιήσουμε και βέβαια η συνθήκη της Λισαβόνας δίνοντας ενιαία νομική προσωπικότητα στην Ένωση είναι πάρα πολύ φυσικό να μας δείχνει το δρόμο για το πώς θα υπάρξει ένα ενιαίο στάτους, συγκεκριμένοι κανόνες και για τα κόμματα και για τα ιδρύματα. Γνωρίζουμε παραδείγματο χάρη μέχρι σήμερα ότι διάφορα ευρωπαϊκά κόμματα έχουν αναμειχθεί στις εκλογές στα κράτη-μέλη. Δεν έχει κανείς ασχοληθεί με το θέμα αυτό ούτε έχει στραφεί καμία χώρα εναντίον των υπαρχόντων σήμερα ευρωπαϊκών κομμάτων. Όμως θα μπορούσε να γίνει με το νομικό καθεστώς που έχουν σήμερα. Δηλαδή χωρίς νομικό καθεστώς. Διότι περί αυτού πρόκειται στην πραγματικότητα. Σημειώνω ότι η πρόταση ε, της Επιτροπής έχει προβεί σε όλες τις προβλέψεις που χρειάζεται να υπάρχουν και που αφορούν στη σχέση με την υπηκουλικότητα ή την αναλογικότητα, τα ζητήματα που έχουν σχέση με την ευελιξία και βέβαια το γεγονός ότι πάμε στις εκλογές του 2014 και πρέπει να πάμε πιο συναρθρωμένοι και πιο ε, προετοιμασμένοι για τις εκλογές αυτές. Επίσης θα δώσουμε απάντηση και λύση μέσω του καθεστώτος αυτού και σε ορισμένα ζητήματα που έχουν κατά καιρού υπάρξει δηλαδή ε, να χρηματοδοτείται ένα κόμμα εφόσον υπάρχουν οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις είτε από τα κόμματα που αποτελείται ένα κόμμα και αυτό αφορά και στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες όπου υπάρχουν περιφέρειες με εκλεγμένα συστήματα, κοινοβούλια και τοπικές κυβερνήσεις, ε, είτε ε, στα ίδια τα κράτη-μέλη, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει πολλές, ε, πολλοί προβληματισμοί γύρω από το πόσα ιδρύματα έχει το κάθε κόμμα, γύρω από ζητήματα που έχουν σχέση με την ύπαρξη πολιτικών γκρουπ μέσα στο κοινοβούλιο και διπλών πολιτικών ομάδων εκτός κοινοβουλίου και τα λοιπά, Όπως αντιλαμβάνεστε η ασάφεια, η νομική ασάφεια επιτρέπει και αφήνει πολλά περιθώρια να γίνουν και λάθη και βέβαια δεν θα ήταν σωστό σε μια εποχή ε, ανόδου του ευρωσκεπτικισμού και οικονομικής κρίσης και προβλημάτων στην Ευρώπη να παρουσιαστούν τέτοια θέματα με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα όπως έχουν σήμερα που να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και σε αυτά τα κόμματα. Γιατί πιστεύω ότι ε, η στάση των πολιτών για τα ευρωπαϊκά κόμματα έτσι όπως τα γνωρίζουν μέχρι σήμερα είναι μάλλον θετική μάλλον αισθάνονται ασφάλεια οι πολίτες οι οποίοι είναι και μέλη των εθνικών κομμάτων να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κόμμα όπου εκεί συνδέονται οι αντιλήψεις ε, τα στελέχη συμμερίζονται τις ίδιες αξίες και αρχές. Και φυσικά σημειώνω με μεγάλη ένταση αυτό που είπε ο Επίτροπος ότι έχει σημασία τα κόμματα αυτά να συμμερίζονται τις αρχές και τις αξίες της Ένωσης και για να υπάρχουν υπό την έννοια των ευρωπαϊκών κομμάτων και για να χρηματοδοτηθούν. Δεν θέλω να προσθέσω περισσότερα κύριε Πρόεδρε στην πρώτη αυτή συζήτηση. Ε, θέλω να τονίσω μόνο ότι μας χρειάζεται ένα νομικό καθεστώς επί τη βάση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο οποίο θα συμφωνήσει και το Συμβούλιο που θα είναι ένα sui generis νομικό καθεστώς που θα συνάδει και θα αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες της Ένωσης, χωρίς να έρχεται σε αντίθεση με τους νόμους των διαφόρων χωρών ή με το σύνταγμά τους. Άρα χρειάζεται αρκετή δουλειά και προς την πλευρά του Συμβουλίου, όπως είπατε κύριε Επίτροπε, και θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω γιατί η Επιτροπή ε, στάθηκε φερέγγια και κράτησε το λόγο της να εντάξει μέσα στο πρόγραμμα του 12 μια ουσιαστική πρόταση για το ευρωπαϊκό καθεστώς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γιαννάκου και θα δώσω τώρα το λόγο στην ε, συνάδελφο Γκερέρο, ο οποίος είναι ο εισηγητής μας για το δημοσιονομικό κανονισμό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε και τον κύριο Επίτροπο. Θα ευχαριστούμε που ήρθε και μας παρουσίασε αυτές τις ε, δύο Τέλο τέλος πάντων την πρότασή του. Όπως είπε και η κυρία Γιαννάκου και εγώ συμφωνώ ότι το Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα η Επιτροπή μας θα πρέπει να είμαι θα ε, ευγνώμονες που μπορέσαμε έτσι να περάσουμε τις προτάσεις μας, τις προτάσεις κυρίας Γιαννάκου και επομένως η ουσία μεταφέρθηκε στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει να προσέξω τον κίνδυνο που ελοχεύει για μένα γιατί εγώ είμαι ο εισηγητής για τον δημοσιονομικό κανονισμό και θα πρέπει να προσέξω μήπως φανεί ότι είναι η ειδική συνταγματολόγος κύριε Γιαννάκου και εγώ ότι είμαι ένας απλός λογιστής. Τέλος πάντων, πέρα από αυτά θα πρέπει επομένω να σας πω δύο πράγματα πέραν επομένως του ρόλου μου ω λογιστή και να σας πω τη γνώμη μου γενικότερα γιατί έτσι κι αλλιώ θα πρέπει συνολικά και συλλογικά να δουλέψουμε. Και ε, δανείζομαι λοιπόν αυτή τη σκέψη που μα διατύπωσε η κυρία Γιαννάκου, ότι δηλαδή θα πρέπει να αναβαθμίσουμε, να ενισχύσουμε την Επιτροπή μα σε σχέση με το, το, το, το, το συζητούμενο νομοθέτημα, το οποίο έχει πάρα πολύ σημαντικέ συνέπειε δημοσιονομικέ. Και φυσικά με το κλίμα και τη σημερινή συγκυρία αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα πρέπει να προσέξουμε το ότι η προβληματική συζήτηση ε, θα στραφεί σε σχέση με το, το ότι τα πολιτικά κόμματα ζητάνε λεφτά, περισσότερα λεφτά και επομένω. επομένως η δική μας θέση και η δική μας νομιμοποίηση θα δεχθεί σημαντικό πλήγμα. Οπότε με κάποιες λίγες ε, εξαιρέσεις πάρα πολύ σεβαστές και θεμητές όμως που δεν αποτελούν τον κανόνα αλλά εξαιρέσεις όλοι οι υπόλοιποι συμφωνούμε ότι σήμερα η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Όλα αυτά τα οποία περάσαμε την τελευταία τριετία είναι κάτι το οποίο κατατείνει προς αυτή την κατεύθυνση προς την διακυβερνητική εκδοχή και θα έχουμε αντιπαράθεση επομένως απόψεων αντιπαράθεση με τόπο βορρά νότου ε, χωρών τριών α και χωρών προβληματικών οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τα οράματα τις ιδεολογίες που έχουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι θέλει ο καθένας για την Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θέλει να είναι η Ένωση σήμερα και στο μέλλον. Οπότε θα πρέπει να μην υπονομεύσουμε αυτή την πολεμική, αυτή την προβληματική. Οπότε αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να έχουμε κατά κάποιο τρόπο κοινό μέτωπο. Σε σχέση με το τι ζητάμε για τα ευρωπαϊκά πολιτικό κόμματα και γι' αυτό πιστεύω πως ε, η πρόταση όχι μόνο ήρθε τη σωστή στιγμή, αλλά είναι και πάρα πολύ εύστοχη. Ήρθε κάποια στιγμή κατά την οποία οφείλουμε να περιχαρακώσουμε, να ενισχύσουμε, να θωρακίσουμε αυτές μας τις ε, ε, απόψεις για τις ευρωπαϊκές εκλογές κατά τις οποίες πέραν των εσωτερικών αντιπαραθέσεων οι πολίτες θα τοποθετηθούν όσον αφορά συνολικά τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα χρηματοδοτικά ακόμη Περιμένουμε την ε, δημοσίευση των διατάξεων που θα διέπουν την χρηματοδότηση και έτσι να μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε τις τροπολογίες μας και να τις υποβάλλουμε. Όπως είπα όμως ε, στην αρχή, αυτές οι τροπολογίες αφορούν κυρίως τα διαδικαστικά ζητήματα της χρηματοδότησης δικαιολόγηση δαπανών, ε, κατανομή των πόρων, πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Όμως, και ας είμαι εγώ εισηγητής, δεν είναι αυτά η ουσία των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό και λέω ότι θα πρέπει να κάτσουμε και να προβληματιστούμε για το σύνολο της πρότασης. Ακριβώς όπως έκανε και η κυρία Γιαννάκου. Δεν θα πρέπει να είμαστε ε, πάρα πολύ σχολαστική δεδομένου του χρονοδιαγράμματο που έχουμε. Και, κύριε Επίτροπε, υπάρχουν κάποια ερωτήματα προς εμάς. Υπάρχει και κάποια αμφιβολία. Αυτό το καταστατικό που θα διέπει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα είναι το μοναδικό νομοθέτημα που θα τα διέπει ή θα πρέπει επικουρικά να έχουμε και κάποια άλλα νομοθετήματα και να συνδυάζουμε αυτό το καταστατικό με κάποια άλλα νομοθετήματα ανάλογα με το που είναι η έδρα του εκάστου πολιτικού κόμματος. Βρυξέλλες, στο Βέλγιο ή κάπου αλλού. Και αν θα συντρέχουν επομένω και οι εθνικές νομοθεσίες. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε διτή πορεία, διπλή δουλειά. Πρώτα-πρώτα να προωθήσουμε νομοθεσία η οποία θα καλύπτει σε ευρωπαϊκό επίπεδο όλα τα νομικά ζητήματα που θα διέπουν τη χρηματοδότηση των κομμάτων και έτσι να το κάνουμε αυτό να μην καταλήξουμε σε μια πολυνομία γιατί έτσι θα προκύψει και σύγχυση και προστριβή και αντιπαράθεση. Δεύτερο ερώτημα το οποίο αναδύεται και σας το υποβάλλω. Τι είδους έλεγχο θα, θα, θα, θα, ασκεί κανείς σε κάποιο πολιτικό κόμμα για το αν αυτό το κόμμα πληρεί τις προϋποθέσεις των ε, αξιών που είπατε. Επί τη βάση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακούμε ότι θα πρέπει το κοινοβούλιο να αποφασίσει εάν δεν συντρέχει περίπτωση τήρηση αυτών των αξιών από κάποιο κόμμα. Και θα γίνει εξολόγηση από τρεις προσωπικότητες που θα προτείνονται από τα τρία θεσμικά όργανα Κομισιόν, Συμβουλίο, Κοινοβούλιο. Να δούμε τι, τι ισχύει όσον αφορά εναλλακτικέ λύσει. Τελικά το Κοινοβούλιο είναι πολιτικό όργανο. Άρα θα πρέπει τελική απόφαση σχετικά με το εάν ένα πολιτικό κόμμα ευρωπαϊκό δεν πληρεί την προϋπόθεση των ε, ευρωπαϊκών αξιών, θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο αυτό να κρίνεται από κάποιο συγκεκριμένο ειδικό όργανο το οποίο εξορισμού θα πρέπει να συγκροτείται με πολιτικά κριτήρια. και εγώ και η πολιτική μου ομάδα δεν θέλουμε πάνω σε αυτό να θεωρήσουμε ότι έχουμε κάποιο συμφέρον, αλλά θα πρέπει να δούμε το αν υπάρχει προηγούμενο σε εθνικό επίπεδο για το αν επομένω ε, αναγνωρίζεται κάποιο φορέα ανάλογα με το αν πληρεί κάποιε τέτοιε αξιακέ προποθέσει. Δεν έχω επομένω καμία ένσταση για το ποιο θα ασκεί αυτόν τον έλεγχο. Όμω θα πρέπει αυτό να ρυθμιστεί πολύ πολύ συγκεκριμένα και να δούμε κατά πόσο θα μπορεί εκ των υστέρων το Κοινοβούλιο με κάποιο πολιτική ψηφοφορία να ανατρέψει κάποια αξιολόγηση στην οποία έχουν προβεί προηγουμένω αυτέ οι τρει ε, προσωπικότητε, εκπρόσωποι των ε, ε, θεσμικών οργάνων. Τώρα, για κάποια άλλα θέματα χρηματοδότηση. Το βασικό θέμα για το οποίο συμφωνώ και είναι πάρα πολύ συμφωνώ ή θα πρέπει να ισχύσουν οι κανόνες της διαφάνειας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι θα αποφύγουμε προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με τη χρηματοδότηση και δεν είναι θέμα αυστηρής ε, ρύθμισης. Είναι το ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Και έτσι ε, έχουν άλλη έννοια οι ιδιωτικές δωρεές και πάσα μορφή χρηματοδότηση. Η πολιτική μου ομάδα έχει ασχοληθεί με δύο θεματάκια τα οποία όμως θέλει κάπως να μεταβάλει. Πρώτα πρώτα, το πώς θα γίνει η κατανομή της χρηματοδότησης. Η σημερινή σας πρόταση λέει ότι το 15% του συνόλου θα πρέπει να κατανέμεται εξίσου εις τα ευρωπαϊκά κόμματα και το 85% αναλογικά με τον αριθμό των μελών που το κάθε κόμμα έχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η κατανομή κατά τη γνώμη μου δεν είναι πιο δόκιμη. Το 15% είναι πολύ που να πηγαίνει δηλαδή το ίδιο σε κάποιον που έχει 200 ευρωβουλευτές και το ίδιο να πηγαίνει σε κόμμα που έχει έναν. Οπότε, να υπάρχει ποσοστό ποσού που να πηγαίνει παντού. Αλλά να μην είναι 15%. Δεν ξέρω πόσο, αλλά να είναι λιγότερο από 15%. Ίσως το 10% να ήταν δικαιότερο. Τώρα, σώμα να την συγχρηματοδότηση. Ξέρετε εδώ πέρα υπάρχουν ποικίλε απόψεις. πολιτική μας ομάδα θεωρεί ότι υπάρχουν ε, κάποιες πολιτικές ομάδες που ελκύουν περισσότερο την ιδιωτική χρηματοδότηση. Περισσότερο από την αριστερά. Περισσότερες δωρεές από ότι οι σοσιαλιστές. Οπότε ε, έχουμε τώρα θέμα υψηλού ποσοστού συγχρηματοδότησης, το οποίο βέβαια δεν θα αρέσει σε κάποια πολιτικά κόμματα. Πάντως ε, αυτό το ποσοστό ξεκίνησε σαν υψηλότερο, τώρα το κατεβάσατε τι προτάσεις σα. Εμείς πάντω θα κατεβάσουμε μια τροπολογία για να έχουμε ακόμα μικρότερο ποσοστό. Επίση συμφωνούμε για ότι θα πρέπει να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία, θα πρέπει να υπάρχουν εκθέσεις ε, κατόπιν των ελέγχων και εν τέλει έχουμε άλλα δύο θέματα στα οποία θέλω να θίξω για να ολοκληρώσω. Πρώτα-πρώτα το θέμα του διαγράμματος Είναι αλήθεια ότι όπως είπε ο κύριος Επίτροπος θα κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς εδώ από το Κοινοβούλιο τόσο ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία της διεκπαιρέωσης. Βέβαια θα φτάσει κάποια στιγμή ο Ιούλιος του 2013 και άρα εκεί έχουμε την καταληκτική ημερομηνία την έχουμε αλλά επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό θα μπορούσε να πάει λίγο παραπίσω να πάει προς το φινόπορο εάν χρειαστεί και αυτό γιατί τα πολιτικά πολιτικόματα χρειάζονται κάποιο χρόνο τόσο ώστε να προσαρμοστούν και να μπορέσουν να συμμορφωθούν προς αυτές τις μεταρρυθμίσεις που κατεβάζετε με την πρότασή σας άλλο ένα θέμα τώρα το οποίο αφορά την αναθεώρηση. Αυτή η προτινόμενη ημερομηνία για την αναθεώρηση λέτε ότι θα πρέπει να γίνεται στο, την τρίτη χρονιά μετά τις ευρωεκλογέ. Αυτό δηλαδή σημαίνει δύο χρόνια πριν την, ε, την διενέργεια των εκλογών. Αλλά ίσως θα πρέπει να είναι στην αρχή της τρίτης χρονιάς την αρχή της τρίτης χρονιάς, ούτως ώστε να υπάρχει περισσότερο χρονικό περιθώριο και για, να, να, να, να αποδώσει αυτή η αναθεώρηση, να, να προκύψει κάτι χρήσιμο ε, και προτάσεις, συστάσεις και κατόπιν ε, ε, αποτελέσματα και έτσι να έχουμε κάποιες μεταρρυθμίσεις για κάποια ζητήματα τα οποία δεν λειτουργούν τόσο καλά. Τώρα για την χρηματοδότηση κάθε αυτή νομίζω ότι η πιο σημαντική επιτυχία θα ήταν να, αυτή η κατάργηση των ετησίων προγραμμάτων και έτσι να είναι πιο ευέλικτη χρηματοδότηση των κομμάτων. Και επίσης να δούμε πώς ε, αυτές οι επιδοτήσεις, οι υποτροφίες, οι χρηματοδοτήσεις να αντικατασταθούν με κάποια εκ των προτέρων δικαιολόγηση ή με κάποια εκ των υστέρων χρηματοδότηση και βέβαια να γίνεται η απορρόφηση και χρησιμοποίηση με ευέλικτο τρόπο. Ευέλικτα και με εύστοχα ε, θεωρούμε ότι είναι αυτά που προτείνεται. Περισσότεροι από εμά εδώ στην Επιτροπή μα, με σεβασμό, με, με, με συμπάθεια βλέπουμε τα όσα προτείνεται και φυσικά και εκτιμούμε το ότι λάβω τη βοήθεια τη προτάσει και αυτό που θα προσπαθήσουμε είναι το να δουλέψουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα για να τηρήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Για ε, εντάξει, να γίνουν και κάποιε αλλαγέ, θα γίνουν από διάφορα πολιτικά κόμματα ε, και φυσικά θα υπάρξουν και κάποιες προτάσεις τροποποιών κόντρα στις δικές μου. Για πέστε μας, πέστε μας το μυστικό. Στο Συμβούλιο, ποιες χώρες αντιστέκονται. Τι γίνεται. Για να μπορέσουμε να πιέσουμε κι εμείς πιο αποτελεσματικά. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Γκερέρο. Δεν έβαλα ε, κανένα χρονικό περιθώριο στην κυρία Γιαννάκου και στον κύριο Γκερέρο γιατί είναι εισηγητέ. Αλλά για να μπορέσουμε να έχουμε την απάντηση ε, του ε, εισηγητού, του, συγγνώμη, για να έχουμε την απάντηση του κυρίου Επιτρόπου θα πρέπει οι παρεμβάσει να είναι πάρα πολύ σύντομε από του συναδέλφου. Τρία λεπτά και πολλά λέω. Κύριε Ντάφ, παρακαλώ. Good Καλησπέρα. Έχω ορισμένε ερωτήσει. Είπατε σωστά ότι υπάρχουν προβλήματα στο Συμβούλιο και πάντα υπάρχουν προβλήματα στο Συμβούλιο. Όμως, ευτυχώς το καταστατικό θα ακολουθήσει τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, δηλαδή ειδική πλειοψηφία. και ελπίζω ότι η Επιτροπή θα επιμείνει να ισχύσει η ειδική πλειοψηφία για να υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα. Δεύτερον, το ότι τα πολιτικά κόμματα πρέπει να είναι καταχωρημένα σε ένα κράτος μέλος και θα υπόκειται σε εθνικό δίκαιο, το οποίο σε αυτά τα θέματα διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί επέλεξε η Επιτροπή αυτή την εναλλακτική λύση και όχι, παραδείγματο χάρη, το να επιτρέπει στα πολιτικά κόμματα να καταχωρούνται με καταστατικό ευρωπαϊκής εταιρείας. Τρίτον, και αυτό είναι πολιτικό σημείο, δεν ε, συμπεριλαμβάνεται τα πολιτικά κόμματα σε εκστρατείες ε, δημοψηφισμάτων, πράγμα που μου, είναι, ε, μου φαίνεται περίεργο, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά δημοψηφίσματα πέραν του κέριου σημείου των ε, αλλαγών στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μου φαίνεται σημείο για το οποίο θα είναι επιθυμητό να παίζουν κάποιο ρόλο τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα σε τέτοιες εκστρατείες. Γιατί απαιτείται μια ευρωπαϊκή διάσταση σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Και επίσης, στην αιτιολογική σκέψη 18 αναφέρεται τη δήλωση της συνθήκης της Νίκαιας για τα πολιτικά κόμματα. Κατά τη γνώμη μου είναι απειχιωμένο αυτό το σημείο και υπάρχει η λειτουργία των πολιτικών κομμάτων ε, στην συνθήκη της Λισαβόνας που είναι περισσότερο σωστή προσέγγιση. Τέλος, ένα διαφορετικό σημείο. Νομίζω ότι η Επιτροπή μας θεωρεί ότι πρέπει να δοκιμαστούν τα πολιτικά κόμματα και να τα υποχρεώσουμε να συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ζητήσουμε λοιπόν από την Επιτροπή να κάνει μία δήλωση στην Ολομέλεια σχετικά με την οργάνωση των εκλογών του 2014 Και στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης θα θέλαμε να καταλήξουμε σε ένα γραπτό ψήφισμα με τρία στοιχεία. Πρώτον, ότι τα πολιτικά κόμματα θα ορίζουν αυτόν που θεωρούν υποψήφιο για πρόεδρο της Επιτροπής. Δεύτερον, ότι 50% των μελών της επόμενης Επιτροπής θα προέρχεται από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τρίτον ότι η ημερομηνία των εκλογών αντί για τον Ιούνιο θα είναι Μάιος. Θα ήθελα τις αντιδράσεις του κ. Επιτρόπου στο θέμα αυτό. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσει και η διάσκεψη των Προέδρων αύριο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχήν ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που έχουν ζητήσει το λόγο και σας παρακαλώ να είστε σύντομοι για να έχουν όλοι ίση μεταχείριση. Ο κύριος Σόλς είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καλώς ήρθατε. Και νομίζω ότι ε, το καθήκον που μας περιμένει για αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Θα μιλήσω με ειλικρίνεια, θα εστιαστώ στα συγκεκριμένα θέματα γιατί έχουμε κάνει μια μεγάλη συζήτηση και τώρα έχουμε ε, το νομοθετικό κομμάτι. Και θέλω να ρωτήσω τα εξής διευρύνεται τον ορισμό των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και συμπεριλαμβάνεται και τα φυσικά πρόσωπα. Ποια είναι η σχέση μεταξύ ενός οργανισμού πολιτικών κομμάτων ε, από κράτη-μέλη έναντι αυτής της έννοιας των φυσικών προσώπων. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα. Και έχουμε την εμπειρία από πολλά πολιτικά κόμματα όταν υπάρχει το θέμα του πώς μπορεί ένα μέλος να επηρεάσει το πολιτικό έργο του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος. Τι δικαιώματα έχει, τι υποχρεώσεις και τι ευκαιρίες συμμετοχής έχει στην διαμόρφωση της δραστηριότητας Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ή και σε άλλες σχετικές δομές. Δεύτερη ερώτηση. Ποια είναι η σχέση μεταξύ εθνικών κομμάτων που είναι μέλη Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος. Διότι αν δείτε τώρα την Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, και σήμερα ένα εξέχον μέλος του ΕΛΚ θα βρίσκεται στην Ελλάδα. Και υπάρχει και μια διαδικασία και με κόμματα άλλων πολιτικών οικογενειών. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό για την ευρωπαϊκή συζήτηση γενικότερα. Πρέπει να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων. Και τρίτον, για τη χρηματοδότηση δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο για μένα. Το γιατί συγχαίρεται την αναγνώριση ως ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, ευρωπαϊκή νομική οντότητα και την αναγνώριση σε ένα από τα κράτη-μέλη. Διότι αυτό δημιουργεί ένα μείγμα ε, στα πρακτικά θέματα των κομμάτων. Παραδείγματο χάρη, τα άτομα που απασχολούνται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα τότε θα υπάγονται στον κανονισμό βάσει στα κράτη-μέλη και όχι στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το μείγμα θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Άγνιου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πραγματικά σύντομος για να κερδίσετε χρόνο από τη δική μου παρέμβαση. Κύριε Επίτροπε, ακούγοντας την πρότασή σας για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, συχνά αναφερθήκατε σε προϋπολογισμό και χρηματοδότηση. Άκουσα από τον συνάδελφο Άντριου Νταφ που σας ζήτησε να χρησιμοποιούνται, να επιτρέψετε να χρησιμοποιούνται αυτά τα κονδύλια για να επηρεάζονται εκστρατείε δημοψηφισμάτων. Στη χώρα μου ιδιαίτερα θα μπορούσε αυτό να γίνει για τις μελλοντικές μας σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ σας παρακαλώ να κάνετε το αντίθετο. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το κάνετε και θα ήθελα τη διασφάλισή σας κατηγορηματικά ότι ποτέ δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Δεύτερον, στα πολιτικά αυτά κόμματα θα πάνε αρκετά, ε, αρκετά χρήματα των φορολογουμένων. Γνωρίζετε ε, να υπάρχει πρώτερη δήλωση κάποιων που έχουν πει ότι θέλουν να χρηματοδοτούν τα πολιτικά κόμματα, ούτε ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε δεν σας πήρα. Μπράβο, μπράβο. α, Άξιος. Ελπίζω και οι άλλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας. Μπρόντς. Ευχαριστώ. Εγώ δεν είμαι υπέρ τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων ούτε από κράτη ούτε από διεθνεί οργανισμού. Θα μπούμε στη φασαρία ε, του ε, ε, να κάνουμε πράγματα που θα πρέπει να κάνουν μόνοι τους. Υπάρχουν όμως δωρές μεγάλης κλίμακας από εταιρείε, από συνδικάτα, από κυβερνήσεις και δεν είμαι υπέρ της χρηματοδότησης ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων διότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ακόμη λιγότερο δεν μπορούν να προσελκύσουν βουλευτές και χρηματοδότηση. Δεν θέλουμε λοιπόν να χρηματοδοτούμε ένα οργανισμό που δεν θα έχει καμία πραγματικότητα. Εάν κάποια κόμματα όμω παίρνουν χρηματοδότηση, θα πρέπει όλα να παίρνουν, διότι δεν μπορεί να χρηματοδοτούνται κάποια κόμματα και κάποια άλλα να μην χρηματοδοτούνται και εδώ υπάρχουν δύο κανόνε. Πρώτον, ότι πρέπει να ισχύουν οι όλοι, οι ίδιοι κανόνες για όλα τα κόμματα, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Και δεύτερον, οι δεν θα πρέπει να εφεύρουμε κανόνες που θα αφήνουν απ' έξω κάποια κόμματα λόγω της πολιτικής τους ή της ιδεολογίας τους. Διαφορετικά τα μεγάλα κόμματα θα μοιράζονται την πίτα μόνα τους και θα απορρίπτουν όλα τα μικρότερα κόμματα. Από την έκθεση της εισηγητήρας φαίνεται ότι τα κόμματα θα πρέπει να έχουν υψηλά πρότυπα διαφάνειας ε, και αξιοπιστίας και δεν νομίζω σε αυτό έχουμε καμιά αντίρρηση, κανείς δεν έχει αντίρρηση. Δεύτερον, θα πρέπει να σέβονται τις αξίες ε, επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι περισσότερε από τι αξίε αυτέ φαίνεται να είναι παγκόσμιε αξίε και φαίνεται να είναι αποδεκτέ, αλλά όχι η ερμηνεία την οποία πολλέ φορέ κάνουμε για αυτέ τι αξίε. Παρότι η ευρωπαϊκή πολιτική τάξη μπορεί να θεωρεί ότι η ερμηνεία τη είναι προφανή και αυταπόδεικτη, φοβούμε ότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι οι δικέ του αξίε είναι πάντοτε αυτονόητε και αυταποδεκτε. αλλά οι αξίε εξορισμού είναι υποκειμενικέ. Ε, οι αξίε είναι υποκειμενικέ κρίσεις. Και τα υποκειμενικά κριτήρια δεν θα πρέπει να έχουν θέση σε νομικά κείμενα. Λοιπόν, οι νομοθετικέ διατάξει θα πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, θα πρέπει να σέβονται το πνεύμα και το γράμμα του κράτου δικαίου. Και τέλο, προτάθηκε νωρίτερα, η τελική απόφαση για το αν ένα πολιτικό κόμμα θα παίρνει χρηματοδότηση να επαφείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το θεσμικό όργανο που είναι το λιγότερο ενδεδειγμένο να παίρνει τέτοια απόφαση, διότι εδώ υπάρχουν κόμματα που έχουν ένομο συμφέρον για τη δική του χρηματοδότηση και ένομο συμφέρον εναντίον όποιων άλλων είναι αντιπαλή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χέφνερ, πάντα να σας ζητήσω να είσαστε σύντομοι, έτσι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ε χαίρομαι που συζητάμε αυτό το θέμα το θεωρώ πολύ σημαντικό, το θεωρώ πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση για μια ευρωπαϊκή δημοκρατία που θα λειτουργεί ακόμη καλύτερα και θα υπάρχει ακόμη καλύτερη αντιπαράθεση διαφορετικών πολιτικών προγραμμάτων και πολιτικών περιεχομένων και κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια ενίσχυση της ζωής μέσα στα πολιτικά κόμματα και μια καλύτερη παρουσίαση των κομμάτων ε, ούτως ώστε ε, οι πολίτες να αντιλαμβάνονται καλύτερα τα πολιτικά κόμματα και να μπορούν να συμμετέχουν καλύτερα και αυτό και μέσω τη διαδικασία των ευρωπαϊκών εκλογών. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον ε, Επίτροπο και την Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Σεύκοβης και να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια την κυρία Γιαννάκου. Ε, Ιδίω είναι σημαντικό αυτό ότι θα υπάρχει νομική προσωπικότητα για τα πολιτικά κόμματα και για τα πολιτικά ιδρύματα. Εδώ υπάρχουν ε, πολλές συνέπειες στην πράξη όσον αφορά και τη χρηματοδότηση. Δεν θα είναι χρηματοδότηση ε, υπό τη μορφή επιδότησης λειτουργίας αλλά υπό τη μορφή συνεισφορών. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις ε, θίγοντας κάποια θέματα τα οποία θεωρώ σημαντικά. Πρώτον, Όσον αφορά τα κριτήρια, πιστεύω ότι είναι σωστό να έχουμε κριτήρια βάση του προγράμματος, του καταστατικού και της εσωτερικής δημοκρατικής τάξης των κομμάτων. Είναι λογικό να έχουμε τέτοια κριτήρια. Αλλά η παρουσίαση ε, υποψηφίων ε, είναι θέμα του κάθε κόμματος και γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω και δεν το θεωρώ και σωστό το να υπάρχει απέτηση ε, δημοκρατικής εκλογής στο άρθρο 4 παράγραφος 2 μικρό δέλτα ότι θα βασίζεται μόνο από τα όργανα καθοδήγησης του κόμματος και όχι από τους υποψηφίους. Νομίζω ότι υπό την έννοια της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας δεν ε, θα έπρεπε να έχουμε ε, υποψηφίου που δεν θα προέρχονται από τη δημοκρατική διαδικασία μέσα στα κόμματά τους και σκέφτομαι και τα κόμματα στις ευρωπαϊκές εκλογές. Τα ευρωπαϊκά κόμματα πρέπει να ζητούν η εσωτερική δημοκρατική τάξη να ισχύει. Δεύτερο σημείο, όσον αφορά τα δημοψηφίσματα που αναφέρθηκε ήδη αυτό το θέμα, νομίζω ότι θα ήταν σημαντικό σφάλμα να αποκλείσουμε εδώ κάποια κόμματα. Τα κόμματα δεν είναι μόνο εκλογικές ε, συσσωματώσεις είναι όργανα διαμόρφωσης και που προέρχονται από την κοινή γνώμη και από την κοινωνία και θα πρέπει να μην ξεχνάμε τα πολιτικά κόμματα ε, στα δημοψηφίσματα, θα πρέπει ενεργά να συμμετέχουν και να τα συμπεριλάβουμε στη διαδικασία. Το επόμενο σημείο τώρα για το οποίο επίσης πρέπει να πω ότι το θεωρώ σημαντικό τα κριτήρια για την ε, χορήγηση άδεια δεν θα πρέπει να είναι τόσο υψηλά όσο για τη χρηματοδότηση. Ε, ε, στην πράξη όμως νομίζω ότι τα κριτήρια για την έγκριση ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων είναι πολύ ψηλά και δεν θα πρέπει να συνδέονται με το επίπεδο της εκπροσώπησης στα εθνικά κράτη ή στο κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε ανταγωνισμό, χρειαζόμαστε νέα κόμματα και γι' αυτό η διαμόρφωση πολιτικών προγραμμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη θα πρέπει να μας ενδιαφέρει άμεσα. Δεν θα πρέπει δηλαδή, να βασίζεται μόνο από τις έδρες που κατέχει ένα κόμμα στο κοινοβούλιο στη χρηματοδότηση θα πρέπει να δούμε ποια κριτήρια θα ισχύσουν. Ξέρω ότι έχω ξεπεράσει το χρόνο μου ή μόλις ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. κύριε κύριος Βίλαντερ και μετά να απαντήσει ο Επιτροπός. Ευχαριστώ αυτό, για, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, ε, θα συνεχίσω μετά από αυτά που είπε ο κ. Χέφνερ, ιδίω όσον αφορά ε, την ε, ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και τους πολίτες και την ισχύ των κομμάτων. Στο άρθρο 3, το 3% στο 1 τέταρτο των κρατών μελών θεωρώ ότι είναι πολύ υψηλό. Νομίζω ότι θα έπρεπε να το αντικαταστήσουμε αυτό με μεγαλύτερο αριθμό χωρών στις οποίες ε, θα πρέπει ε, να συμμετέχει το κόμμα ενεργά στις ευρωπαϊκές εκλογές. Θέλουμε να εκπροσωπείται το κόμμα στις ευρωπαϊκές εκλογές και αυτό θα είναι σημαντικό ε, για ένα κόμμα και για το καταστατικό του. Και θα θέλουμε να έχει απήχηση ένα κόμμα στις, στις εκλογές. Μετά στο άρθρο 5 μιλάμε για νομικά πρόσωπα τα οποία μπορούν να είναι μέλη των κομμάτων. Όταν ένα κόμμα λέει ότι ε, ε, για μας θα είναι μέλη όλα τα μέλη της ε, ΕΛΠΑ, τέλος πάντων της ε, Λέσχης Αυτοκινήτου, θα είναι όλα τα μέλη της ΕΛΠΑ, μέλη του κόμματος. Θα πρέπει να δούμε ε, ποια είναι τα πραγματικά πρόσωπα, τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη των κομμάτων και για λόγους εκπροσώπησης νομίζω θα πρέπει να μιλάμε για συμμετοχή στα κόμματα και στα ανώτερα επίπεδα θα πρέπει να επιλέγονται με ε, μυστική ψηφοφορία και νομίζω θα πρέπει να ισχύσουν όλες οι δημοκρατικές επιταγές για τα πολιτικά κόμματα. Επίσης είναι σημαντικό η πρόσβαση σε υποψηφιότητα να είναι εφικτή και θα πρέπει να είναι σαφές ότι οι εκπρόσωποι ε, θα έχουν ίσα δικαιώματα, κάθε μέλος δηλαδή μπορεί να έχει ε, ίσα δικαιώματα στις δημοκρατικές εκλογές και εδώ θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις υποψηφιότητες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να ζητούμε την μυστική ψηφοφορία για την επιλογή των υποψηφίων. Πολλοί λένε ότι η μυστική ψηφοφορία δεν θα πρέπει να ισχύσει γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια. Ξέρω ότι υπάρχει αυτό το επιχείρημα. Τώρα το 85% θα πρέπει να δούμε ε, τι είναι. Μπορεί να μετράμε μόνο τα μέλη τα οποία είναι εκλεγμένα στο Κοινοβούλιο και εκπροσωπούνται λόγω δημοκρατικής ψηφοφορίας από τους ε, ψηφοφόρους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Γκουρμάη. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που καθυστέρησα να έρθω, αλλά ε, είχαμε τη θεσμική ομάδα για την πληροφόρηση όπου αντικαθιστούσα τον πρόεδρο Κασίνη. Θα ήθελα ε, να καλωσορίσω τον αντιπρόεδρο κ. Σεύκοβιτς. Σας ευχαριστώ για την ε, παρουσία σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια την κυρία Γιαννάκου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί Κοιτά αυτό το καταστατικό εδώ και πολύ καιρό και χαίρομαι ιδιαίτερως που καταφέραμε τελικά να δουλέψουμε πάνω σε αυτή την πρόταση κανονισμού για το καθεστώς χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, γιατί και αυτό το θεωρώ σημαντικό. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα από πολιτική και από δημοκρατική πλευράς, ιδίω καθοδόν προ τι επόμενε ευρωπαϊκέ εκλογέ. Η νομική προσωπικότητα την οποία θα έχουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα θα βελτιώσει την πολιτική αναγνώριση. Θέλουμε να τονίσουμε τη δημοκρατία και γι' αυτό τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητα. Χρειάζονται το σωστό πλαίσιο για να εκπληρώσουν το ρόλο τους όπως προβλέπεται στις συνθήκες και αυτό θα βελτιώσει και την διαφάνεια και την δυνατότητα ελέγχου ιδίω όσον αφορά και την τήρηση των ευρωπαϊκών αξιών. Σε μια περίοδο που οι Ευρωπαίοι πολίτε νιώθουν απόμακρα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αυτή την εποχή που υπάρχει τόση ανησυχία για τα όσα γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πιστεύω ότι έχει εξαιρετική σημασία το να ενισχύσουμε τα ευρωπαϊκά κόμματα. Είναι μια πραγματική ευρωπαϊκή συζήτηση και θα πρέπει οι φωνέ των πολιτών ε, να ενωθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδίω σε εποχέ κρίση ε, υπάρχει και δημοκρατικό έλλειμμα και η ενίσχυση των ευρωπαϊκών κομμάτων τελικά θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατά τρόπο δημοκρατικό και διαφανή. Ε, πρακτικά τώρα υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που θα πρέπει να λύσουμε το το κατά πόσο είναι εφικτό το διπλό νομικό καθεστώ. Πάντως ε, χαίρομαι που περάσαμε σε αυτό το στάδιο και θα προσβλέπω σε μια πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο ε, κύριε ε, τον κύριο Σεύκοβιτς. Ευχαριστώ εκ των πρωτών του διερμηνείς γιατί θα μείνουν λίγο ακόμα μαζί μας, 10-15 λεπτάκια. Ε, ε, τους ευχαριστώ εκ των προτέρων λοιπόν και δίνω το λόγο αμέσως στον Πρόεδρο Σεύκοβιτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους ε, για τα σχόλια και θα ήθελα να σας απαντήσω. Νομίζω λοιπόν ότι και η κυρία Γιαννάκου αλλά και ο κύριος Ενρίκε ε, Γκερέρο και η κυρία Γκουρμάη είναι μια εξαιρετική ομάδα για να δουλέψει για αυτό το θέμα ε, και το είδαμε και στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο όλα είναι μια εξαιρετική ε, ομάδα όλα αυτά που μας είπαν είναι πάρα πολύ σημαντικά πιστεύουμε ότι η πρόταση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα να να φτάσουν σε ένα ίδιο καθεστώς και ίδιο επίπεδο τα ευρωπαϊκά ε, πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα ε, γιατί αυτό που προσπαθούμε είναι ε, να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο και όσον αφορά τη χρηματοδότηση και όσον αφορά τη διαφάνεια θέλουμε να γίνουν πιο σαφείς οι κανόνες, να γίνει πιο διαφανής η άντληση χρηματοδοτήσεων κτλ. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε την Ένα ε, ε, sui generis νομοθετικό ε, πλαίσιο για την αναγνώριση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ήδη έχει πάρα πολύ μεγάλη πολιτική σημασία και πολιτικό βάρος. Πρέπει να υπάρχει σαφήνεια όσον αφορά το, την θέση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων στον ευρωπαϊκό πολιτικό ορίζοντα. Ο κύριος ε, Γκερέρο αναφέρθηκε εν λεπτομερία σε διάφορα στοιχεία ε, των ε, δημοσιονομικών πτυχών της πρότασης όταν ο δημοσιονομικός κανονισμός θα έχει εγκριθεί, τότε θα γίνει και η συγκεκριμένη πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι σε θέση να παρουσιάσει την τροποποιητική ε, πρόταση επί του δημοσιονομικού κανονισμού ε, και εκεί θα μιλήσουμε για, τον οικονομικό και ε, τον, για το οικονομικό και νομικό καθεστώς της, του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος. Βεβαίως ε, θα πρέπει να αποφευχθεί το λεγόμενο double legal status. Ε, θέλουμε να αποφύγουμε το ενδεχόμενο αυτό, τη δυνατότητα αυτή, γιατί αφού έχουν καταγραφεί τα κόμματα σαν ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, τότε έχουν το ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς. Αυτό θέλουμε να έχουμε μόνο. Βεβαίως ε, τα κράτη-μέλη πρέπει να στηρίξουν γιατί βλέπουμε ότι θα χρειαστεί αυτό που εγώ ονομάζω ελαφρά ενσωμάτωση ε, έτσι ώστε ε, σε θέματα εργατικού νόμου, σε θέματα ε, φορολογικού καθεστώτος. Ίσως θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες ε, ενσωματώσεις και προσαρμογές. Εμείς θελήσαμε να ακολουθήσαμε την οδό αυτή γιατί ξέρουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα οδηγήσει τελικά σε μια ενιαία αντιμετώπιση και επομένως θα οδηγήσει και σε εναρμόνιση νόμων, πλαισίων ε, κτλ. Μια ελαφρά λοιπόν ε, ενσωμάτωση όπως την ήπια ενσωμάτωση όπως την ονομάζω εγώ που ευελπιστώ ότι ε, μέχρι, τον επόμενο, ε, το επόμενο καλοκαίρι θα έχουν λυθεί όλα αυτά τα ζητήματα. δύο μιλητές σημείωσαν πόσο σημαντικό είναι το θέμα της διαφάνειας. Βεβαίως το θεωρούμε και εμείς εξαιρετικά σημαντικό. Γι' αυτό λοιπόν δίνουμε μεγάλη σημασία στην ε, διαφάνεια. Ειδικά η άντληση χρηματοδοτήσεων θα πρέπει να γίνεται σε απόλυτη διαφάνεια και βεβαίως με σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών. Και ο κύριος Μπρούς και ο κύριος Άγνιου συμφώνησαν ότι αυτό που ανέφερα για τις ευρωπαϊκές αξίες είναι αδιαμφισβήτητο. Πιστεύω ότι αυτές είναι ούτως ή άλλως καθολικές αξίες, είναι οι αξίες επί των οποίων όλα τα πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη θα πρέπει να ε, βασίζουν ε, ε, το πολιτικό τους έργο και βεβαίως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξέρει πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα πράγματα και ξέρουν, ξέρει το Κοινοβούλιο πάρα πολύ καλά ε, πόσο πρέπει να σεβόμαστε αυτές τις καθολικές και παγκόσμιες αξίες. Διαφάνεια στη χρηματοδότηση και στην άντληση χρημάτων νομίζω ότι έχουν αποσαφινιστεί καλύτερα οι κανόνες. Έχουμε τώρα πολύ συγκεκριμένους κανόνες για το ε, μέγιστο ποσοστό χορηγία αναχορηγό, ε, αναδορητή, πώς πρέπει να γίνονται οι προεκλογικές εκστρατείες, πόσο γρήγορα θα πρέπει να ε, αναφέρονται, αναφέρεται η δημιουργία των, του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος, πώς πρέπει να δημοσιεύεται ο κατάλογος των δωρητών χορηγών και πώς ακριβώς γίνεται η άντληση ε, πόρων. Ε, προβλέπουμε την λογοδοσία, προβλέπουμε επίσης τον εκτονιστέρων έλεγχο, ex έλεγχο, έλεγχο και ε, βεβαίως θέλουμε τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να έχουν καλύτερα αποτελέσματα και θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την άντληση χρηματοδοτήσεων γιατί οι κανόνες που διέπουν το σύστημα είναι πολύ καλύτεροι και πολύ πιο σαφής. Δημιουργούμε το νομικό πλαίσιο έτσι ώστε ε, να ε, μην υπάρξουν προβλήματα στο μέλλον. Τώρα πώς θα είναι η γραμμή του προϋπολογισμού, πώς θα ε, προχωρήσει, πώς θα γίνουν οι συζητήσεις, θα το δούμε αυτό. Νομίζω ότι το νομοθετικό πλαίσιο που δημιουργούμε μας δίνει την δυνατότητα να πάμε προς μια κατάσταση όπου όλοι θα ξέρουν πώς έχουν βρεθεί τα χρήματα, πώς έχουν χρησιμοποιηθεί με μεγάλη διαφάνεια. Όσον αφορά τις ανησυχίες του κυρίου Γκερένα για το χρονοδιάγραμμα, πρέπει να πω ότι το Συμβούλιο είχε ήδη τις τέσσερις συζητήσεις ε, για το θέμα αυτό και η τελευταία θα νομίζω θα λάβει η χώρα αυτή την εβδομάδα. Ε, κρίνοντας λοιπόν με, άλλα νομοθετικά, με άλλες νομοθετικές προτάσεις η ταχύτητα είναι γρήγορη. Βεβαίω έχουν προκύψει ερωτήματα, δημιουργούνται κάποιε ομάδε κτλ. Αλλά πιστεύω ότι μέσω της εντατικής διαβούλευσης με την Κομισιόν ε, και την ε, εμπλοκή, την ενεργή εμπλοκή των εισηγητών και των μέλων των ε, αντιστοίχων επιτροπών οπωσδήποτε θα προχωρήσουν τα πράγματα. Και θα ήθελα να καθησυχάσω τον κύριο Νταφ που βλέπει κλασική περίπτωση συναπόφασης ε, πιστεύουμε ε, και εμείς ότι θα πρέπει ε, η απόφαση να λαμβάνεται με ενισχυμένη πλειοψηφία. Έκανε συσχετισμό ο κύριος Ντάφ με το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας, θα το δούμε αυτό, αλλά βεβαίως η Ευρωπαϊκή, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να λειτουργούν σαν μη κερδοσκοπικού σκοπού οργανισμοί. Νομίζω ότι είναι πιο δόκιμο και πιο σωστό να δημιουργήσουμε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Βεβαίως τα θέματα των δημοψηφισμάτων είναι σημαντικά. Γνωρίζετε ότι έχει ήδη συζητηθεί το θέμα εκτενώς και σε πολλές περιπτώσεις. Βεβαίως αντιμετωπίζουμε με μεγάλη προσοχή το ζήτημα αυτό. Και εδώ νομίζω ότι μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα εθνικά δημοψηφίσματα, ακόμα και αυτά που έχουν ευρωπαϊκά θέματα, ξεπερνούν τις ε, δικαιοδοσίες ε, που αποδίδονται από τις ε, συνθήκες και επομένως ξεπερνούν τα σχετικά άρθρα. Όπως είπα, έχει γίνει πολύ μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό και επομένως μόνο οι εξαρτήσεις πληροφόρησης μπορεί να χρηματοδοτούνται και βεβαίως θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να, ε, στηρίζουμε το θέμα αυτό. Από την άλλη πλευρά βέβαια βλέπουμε λίγο, ε, παίρνουμε και το σφιγμό των ε, πολιτικών, συγγνώμη, κρατών μελών, βλέπουμε πώς αντιμετωπίζουν κάποια πράγματα και τα πολιτικά κόμματα. Και τα λαμβάνουμε όλα αυτά και τα συνυπολογίζουμε στην πρότασή μας. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ταφ γιατί μου έστειλε ε, το ψήφισμα, το κείμενο δηλαδή του ψηφίσματος και ε, βεβαίως μια και μιλάτε και για θέματα ε, που αφορούν την επόμενη Κομισιόν θα πρέπει να διαβάσω πολύ προσεκτικά το κείμενό σας, να ξέρω τι με περιμένει. Ε, βεβαίως θα προωθήσω τα ζητήματα αυτά και θα τα συζητήσω και με άλλους συναδέλφους μου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί ακόμα θα γίνει συζήτηση και για αυτό το θέμα. Ο κύριος Χέφνερ έθιξε το θέμα των υποψηφίων. Νομίζω ότι αυτό που θέλαμε να διασφαλίσουμε είναι το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει και εσωτερική δημοκρατία στους, ε, στα κόμματα, δηλαδή ότι θα πρέπει να γίνουν σεβαστοί οι κανόνες ε, εσωτερικής ε, δημοκρατίας. Η εκλογή, ας πούμε, των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων δεν ε, μας αφορά. Το άρθρο 4.2 αφορά μονάχα τις ε, τους διακυβερνητικούς οργανισμούς και όχι τους απλούς ε, υποψηφίους. Βέβαια μπορούμε να το αποσαφηνίσουμε περαιτέρω και να λύσουμε και αυτό το θέμα. και θα είμαστε στη διάθεσή σας. Και ο κύριος Χέφνερ επίσης αναφέρθηκε και την ε, καταχώρηση και την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού, των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων. Είχα πολλές ε, και εκτενείς επαφές και διαβουλεύσεις ε, με το Κοινοβούλιο και μέσα περιπτώσει καταλήξαμε ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μπορούν να καταχωρούνται εάν καλύπτουν τα κριτήρια, αλλά η πρόσβαση στη χρηματοδότηση μπορεί να γίνεται μονάχα στις περιπτώσεις όπου υπάρχει τουλάχιστον ένας εκλεγμένος ε, βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από αυτό το ε, κόμμα. Δηλαδή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποδείξει ότι είναι παρόν στην ε, ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή και ότι εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία θα είναι τελικά αποτρεπτικά για οποιαδήποτε κερδοσκοπικού χαρακτήρα τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού, του κανονισμού της λειτουργίας, ε, αποφυγή απατών ε, κτλ. Αυτό ε, εγώ το είπα για την καταχώρηση, τα υπόλοιπα, γιατί, που θα καταγράφονται δηλαδή, που θα καταχωρούνται. Στην περίπτωση καταχώρησης και εδώ στρέφομαι και προς τους συναδέλφους να με βοηθήσουν, να με διορθώσουν. Εκεί υπάρχουν δύο κριτήρια Πρώτον, 7 πολιτικές προσωπικότητες από 7 χώρες μέλη που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν το Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα ή 7 πολιτικά κόμματα τα οποία ξεπερνούν τουλάχιστον το 3% ε, ε, επέτυχαν 3% τουλάχιστον στις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές και βεβαίως εσείς θα πρέπει να απευθύνετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το αίτημα καταχώρησης ε, και επομένως εάν έχετε καλύψει είτε το ένα είτε τον τον άλλο όρο, τη μία ή την άλλη προϋπόθεση τότε μπορείτε να καταγραφείτε σαν Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα. Ο κύριος Βιλάντερ επίσης ε, αναφέρθηκε σε χρηματοδοτικά θέματα, δημοσιονομικά θέματα, κυρίως όσον αφορά την διαφάνεια που πρέπει, που πρέπει να έχουν τα οικονομικά των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Βέβαια, βεβαίω μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω την αρχική πρόταση και θα το κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος, εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε Σεύκοβιτσε. Πολλές φορές είχαμε ανταλλαγή απόψεων μαζί σας και ήταν κάθε φορά εξαιρετική η ανταλλαγή αυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας υπομείνατε γιατί καθυστερήσαμε να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά. Ε, ε,